So Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να προχωρήσω στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν έχετε αντιρρήσει. Και πριν καλωσορίσω την Ντανιέλ Νουή για να ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχω μια σημαντική ανακοίνωση Αντόλφο Μπαρμπέρα, κεφαλής της γραμματείας μας, απεσπάστη στην ομάδα του Brexit της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, του επικεφαλής διαπραγματευτή, δηλαδή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μουσελ Νταρνιέ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια ξεκινώ λέγοντας. Πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός. Και βεβαίω ελπίζουμε ότι θα βελτιώσει την εξαιρετική ήδη σχέση που έχει το Κοινοβούλιο με την ομάδα του επικεφαλής διπραγματευτή. Έχει αναλάβει διαφορετικούς ρόλους εδώ και 10 χρόνια στην Επιτροπή μας, αρχικά ως διοικητικός τέλεχος, στην ε, συνέχεια ως πρόσωρινος τμήματάρχης, μετά αναλαβες μόνιμα τη θέση του τμήματάρχη και έχεις υπηρετήσει τη γραμματεία και λόγω των ε, πολύ ικανών σου γνώσεων, της διευθυνσιμότητας, των ικανοτήτων σου και μάλιστα σε περιόδους πολύ δύσκολες ε, τα τελευταία χρόνια. Έχεις προσφέρει λοιπόν σημαντική υπηρεσία. Εγώ προσωπικώς που σε γνωρίζω το 2014 δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω και να επιρρώσω περαιτέρω αυτά τα λόγια. Ήταν τιμή λοιπόν και χαρά η συνεργασία μαζί σου. Ήταν εξαιρετική η δουλειά σου ως ε, επικεφαλής της γραμματείας μας, σε συνεργασία και θέλω να σας συγχαρώ για την βοήθεια που μου έχει προσφέρει σε μένα αλλά και σε όλους μας με τον υψηλό επαγγελματισμό που σε διακρίνει. Έχει εργαστεί εντατικά τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Έχει δραματίσει ω εκ τούτου ε, καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ε, ρυθμιστικό τσουνάμι, μπορώ να πω, που οδήγησε τελικά στην ε, σύσταση τη νομοθεσία για τι τράπεζε, την Τραπεζική Ένωση, τον μηχανισμό σταθερότητα. Και έχοντα την τιμή να συνεχίζω να αναλαμβάνω και να διαδέχομαι τη Sharon Bowles, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και αυτή σου την ε, ε συνεισφορά στις προσπάθειές μου ως Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα μας λείψεις λοιπόν. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η παρουσία σου στην ομάδα αυτή του Brexit θα ε, σηματοδοτήσει πολύ σημαντική ε, προστιθέμενη αξία. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά. Και τώρα, βεβαίως, εκφράζοντας τη θλίψη και τα συλληπιτήρια για όλα τα θύματα που είδαμε τις τελευταίες μέρες, πολύ δυσάρεστες μέρες και στον Ρωμανό Βασίλειο και στην Πορτογαλία. Απευθύνουμε λοιπόν θερμά συλληπιτήρια στους ε, οικείους και τα θύματα των ε, καταστροφικών πυρκαγιών του Λονδίνου αλλά και της Πορτογαλίας. Παρακαλώ, Παγμός Πεγές. Ναι, ως πρώην πρόεδρος τη Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα ήθελα και εγώ να, απευθύνω να αποτίσω φοροτιμή στις ε, ικανότητες του Αντόλφο και να επισημάνω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα στη γραμματεία μας επέδειξε όλες αυτές τις ικανότητες που πολύ εύστοχα υπογραμμίσατε. Θα ήθελα ωστόσο ταυτόχρονα και να χαιρετήσω την εκλογή στη Βουλή των Κοινοτήτων της Άννη ε, Ντότζ, η οποία επίσης θα έχει δραστήριο ρόλο και θα είναι ε, χρήσιμη παρουσία της και σε αυτή τη διαπραγμάτευση για το Brexit. Brian Hayes. Ναι, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Αντόλφο για την ε, επιφανή αυτή θέση που αναλαμβάνει στη διαπραγματευτική ομάδα για το Brexit αναγνωρίζοντας την εξαίρετη υπηρεσία που έχει προσφέρει τα τελευταία δέκα χρόνια στην Επιτροπή μας, γιατί εγώ είμαι μέλος μόνο τρία χρόνια στην Επιτροπή, γνωρίζω πόσο σημαντικό ήταν ο ρόλος συνεισφορά του, η συμβολή του στην προεγωγή όλων των ε, θεμάτων και ως ε, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, σε συγχαίρουμε, σε ευχαριστούμε και είμαστε στο πλευρό σου στο δύσκολο αυτό έργο που αναλαμβάνει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε τώρα στη δημόσια κρόαση. Καλωσορίζω, όπως είπα και πριν, την κυρία Ντανιέλ Νουή, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι η πρώτη για το 2017, όπως προβλέπετε από τη Διοργανική Συμφωνία και το, τη Συμφωνία για τον Μηχανισμό. Ε, στις 23 Μαρτίου είχαμε την προηγούμενη συνάντησή μας με την παρουσίαση του της εκθέσεις για το 2016. Ε, είναι εύστοχη η στιγμή αυτής της συνάντησης ε, που έχει τόσο επίκαιρα θέματα και βέβαια θέλουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση όπως έχει εν ώψη ασφαλώς και της πρώτης περίπτωσης εκαθάρισης της ε, Banco Popular στην οποία είχε σαφή συμμετοχή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και βεβαίω θέλουμε να ακούσουμε και τα σχόλιά σας ε, για τη δουλειά που συνεχίζετε, για το πακέτο για τα τραπεζικά και για τα ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια της προτάσεις του ε, Μαρτίου του 2017. Και βέβαια περιμένουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε πάνω απ' όλα τις ε, εκτιμήσεις σας για τις συνέπειες του Brexit και ιδιαίτερα τις σχετικές με το τραπεζικό τομέα. Θα ήθελα πάντως, ξεκινώντας, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία της εκαθάρισης ε, προχώρησε ε, γρήγορα και βέβαια χάρη και στη στάση του αγοραστεί προκειμένου να αποφευχθεί ένα επώδυνο μπέιλιν και μεταφορά των κρίσιμων λειτουργιών της τράπεζας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να επισημάνω ότι με ανησυχεί το γεγονός ότι χρειάστηκε να φτάσουμε στην, στον κίνδυνο της ανακήρυξης μιας τράπεζας ως ε, αφαιρέγγειας ή πιθανώς αφαιρέγγειας για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή της εκαθάρισης και ότι αυτή η τράπεζα είχε περάσει από δύο ε, τεστ αντοχής. Με επιτυχία. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι έχει τη σημασία της η ε, αυτοψία αλλά ε, πάλι είναι ανησυχητικό το γεγονό ότι πριν από την απόφαση για την εκαθάριση τη τράπεζα δεν είχαν ληφθεί άλλε ε, αποφάσει ή ε, προληπτικά μέτρα. Επομένω, ναι, θεωρούμε ότι είναι μια στιγμή σημαντική επιτυχία για το μηχανισμό στήριξη ταυτόχρονα και θα θέλαμε να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια. Επίσης ανησυχίες εκφράζονται λόγω της ε, ατέλειας του πλαισίου μας δεν έχουμε το έντις, δεν έχουμε το μπάνκις, δεν έχουμε το ντεμπρέλ. Θα χρειαστούν χρόνια για να εισαχθούν ε, σε λειτουργία και βεβαίω θα εξαρτώμαστε για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να ταθούν αυτά σε λειτουργία, από την ανάδειξη ιδιωτών αγοραστών. Αν όμως δεν προκύψει ιδιώτης αγοραστής, τι θα συμβεί. Αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες γιατί θα χρειαστεί να μπουν σε λειτουργία τα ε, συστήματα εγγύηση καταθέσεων και αυτό δεν αφορά μόνο την Ισπανία αλλά και την Πορτογαλία ενδεχομένω. Έτσι λοιπόν ε, ε, αντιλαμβανόμαστε πόσο λίγο είναι ο εξοπλισμό, πόσο ανεπαρκή είναι ο εξοπλισμό που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε σημαντικέ τραπεζικέ κρίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας πω καταρχήν πως ε, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι πάρα πολύ και τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Πορτογαλία, όλους όσους περνάνε αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολες στιγμές ε, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν. Θα ήθελα να πω πως χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας μιλήσω για μια σειρά από πολύ επίκαιρα και σημαντικά θέματα για την τραπεζική εποπτεία στην Ευρώπη. Στα εισαγωγικά μου σχόλια θα μιλήσω για την εφαρμογή ε, των υποπτικών διατάξεων και των συνεπειών του Brexit, όπως επίσης και για κάποια πολύ κομβικά ζητήματα στο πακέτο για τη μείωση του κινδύνου, που αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και να σας πω αυτή τη στιγμή τι κάνουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να σας πω πως η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη πρόκληση για την Τραπεζική Ένωση, αλλά επίσης αυτό συγκεντρώνεται σε κάποιες χώρες. Έχουμε μεγάλους όγκους από κόκκινα δάνεια, τα οποία συνεισφέρουν σε χαμηλή κερδοφορία για τις τράπεζες και επίσης οι τράπεζες δεν είναι σε μεγάλη, δεν έχουν ιδιαίτερη ε, δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Εμείς ως επόπτες ε, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων από την αρχή της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Εποπτείας. Το Μάρτιο φέτος μετά από μεγάλες και εκτεταμένες διαβουλεύσεις η ΕΚΤ δημοσίευσε κατευθυντήρες γραμμές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εφαρμόζονται από όλα τα αντίστοιχα ταμεία και τράπεζες και έχει ζητήσει από τις τράπεζες που έχουν υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων να εφαρμόσουν φιλόδοξες και ρίσκες στρατηγικές για να μειώσουν το επίπεδο αυτών. Έτσι λοιπόν σε κάποιες χώρες έχουμε ήδη καλά αποτελέσματα και τους πιο πρόσφατους μήνες είδαμε πως αρκετές τράπεζες άρχισαν το θέμα των περιουσιακών στοιχείων, των στοιχείων ενεργητικών να το αντιμετωπίζουν πολύ πιο δραστήρια. Εμείς με τα υποπτικά μας όργανα και τις υποπτικές ομάδες θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε στενά και τις προκλήσεις αυτές με τα κόκκινα δάνεια και πώς εφαρμόζουν τη στρατηγική. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε κάποιες πιο προχωρημένες λύσεις έτσι ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Μία σημαντική προϋπόθεση για να έχουμε μία μείωση μη εξυπηρετούμενο δανείο και να μην έχουμε τέτοια σώρευση στο μέλλον είναι οι επόπτες να έχουν επαρκής εξουσίως έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι τράπεζες θα κάνουν έγκαιρη προληπτική ε, στρατηγική έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν ε, τις απώλειες από τέτοιου είδους μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίσης έχουμε τονίσει την ανάγκη να ενισχύσουμε το πακέτο το νομοθετικό το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω επίσης πως για τα κόκκινα δάνεια χρειαζόμαστε να είμαστε αποφασιστικοί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι μόνο οι υπόπτες και επιπλέον της δικής μας δουλειά, χρειαζόμαστε μέτρα θεσμικά, νομοθετικά και κυρίως στα θέματα της αφαιρεγιότητας και των διαφόρων δικαστικών, ε, καθαριστικών διαδικασιών. Τώρα, για την προετοιμασία του Brexit που αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των εργοσιών μας να σας πω ότι από το δημοψήφισμα του 2016 η ΕΚΤ προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης. Πρώτα απ' όλα εξασφαλίζουμε πως οι τράπεζες του χώρου του ευρώ και κυρίως αυτές οι οποίες έχουν θεατρικές ή υποκαταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επίσης και αυτές που έχουν άλλου είδους επιχειρηματικούς δεσμούς με τη χώρα, έχουν αυτή τη στιγμή επαρκή σχέδια επίγουσας ανάγκης για να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα ενός σκληρού Brexit. Δεύτερον, στην ΕΚΤ προετοιμαζόμαστε για όλες τις επιχειρημα... επιχειρησιακές α, ε, ε, πτυχές που σχετίζονται με μια πιθανή επανεγκατάσταση με την κατάσταση τραπεζών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, οι τράπεζες οι οποίες θα μετακινηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Τραπεζική Ένωση θα αντιμετωπιστούν με ισότιμο τρόπο ανεξάρτητα από τον τόπο τον οποίο ενδεχομένω θα επιλέξουν και πως δεν θα υπάρχει καθόλου περιθώριο για οποιοδήποτε είδους αρμπιτράζ μεταξύ εποπτικών προσεγγίσεων. Γι' αυτό αυτό θέλουμε να υπάρχει συνεκτική αντιμετώπιση των ιδιωτικών τραπεζών που θα εγκατασταθούν ή θα μετεγκαταστήσουν κάποιε δράσει στην περιοχή του ευρώ. Είναι περιορισμένα τα όσα μπορούμε να κάνουμε και βεβαίω ανησυχούμε. Αλλά οι κανονιστικέ διαφορέ που έχουμε από τι εναλλακτικέ λύσει που έχουν επιλέξει τα ευρωπαϊκά κράτη ε, αυτή τη στιγμή δημιουργούν ανισορροπίες στο πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποιες ε, πτυχές που απαιτούνται του Brexit και επίσης κάποιες τράπεζες που έρχονται στο χώρο του ευρώ μπορεί αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτούν κάποια παραθυράκια εποπτικά γιατί ε, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν παρόμοιες με τραπεζικές δράσεις ή μη τραπεζικές δράσεις μέσω κάποιου επενδυτικού κεφαλαίου ή κάποιων υποκαταστημάτων τρίτης χώρας ή κάποιων χρηματιστικών επενδυτικών, ε, επενδυτικών μη τραπεζικών δράσεων που θα επιλέξουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη τη στιγμή που θα χαράξουμε πολιτική. Αυτή τη στιγμή η, η CRP, CRD ε, αξιολόγηση που γίνεται δίνει στον νομοθέτη τη δυνατότητα να κλείσει τα παραθυράκια, να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση και ένα από τα παραδείγματα είναι η ενδιάμεση μητρική και υποπτική αυτής που αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο έτσι ώστε ή τα υποκαταστήματα τρίτων κρατών των διεθνών ομίλων που εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή εποπτική νομοθεσία να υποπτεύονται καταλήλως. Ένα άλλο θέμα είναι η εποπτεία μεγάλων επενδυτικών εταιριών ε, που δημιουργούν συστημικούς κινδύνους και εδώ είναι κάποιες πολύ περίπλοκες δραστηριότητες που θα πρέπει να υποπτεύονται ε, συνολικά, σφαιρικά, έτσι ώστε να επιτύχουμε τις ουσιαστικές συνέργειες που χρειαζόμαστε όταν ε, κάνουμε αυτή την εποπτεία σε ε, δράσεις στην αγορά τραπεζικές και επενδυτικές ε, σε επίπεδο peer-to-peer. -peer. to peer είναι μια γνωστή πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τα βασικά σημεία της τραπεζικής νομοθεσίας. Θα ήθελα να μιλήσω καταρχήν για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση κινδύνων. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θα είμαι λοιπόν πολύ ε, σύντομη. Θα μιλήσω καταρχήν πρώτα για τα όσα συμφωνήσαμε έτσι ώστε να έχουμε fast track διατάξεις για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και θα πρέπει να έχουμε ένα αρχικό ε, phasing in με μια ε, εύκολη στρατηγική έτσι ώστε να πετύχουμε το ε, CET 1, δηλαδή το Common Equity Tier 1, που είναι ο λόγος κεφαλαίου υποχρεώσεων κεφαλαίου κοινών μεσών της κατηγορίας 1, έτσι ώστε οι ενδιάμεσες διατάξεις να είναι αρκετά περίπλοκες ώστε να καλύψουν όλα τα σενάρια. Επίσης αυτή η προσέγγιση θα πρέπει de facto να αναβάλει τη θέση σε εφαρμογή του πλαισίου ε, διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 9, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να υπολογίζουμε τις διατάξεις και να δούμε ποια είναι τα επίπεδα κεφαλαίου και επάρκειας κεφαλαίου που θα έχουν οι τράπεζες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις CET1 για να καλύψουμε όλη την ενδιάμεση περίοδο. Δεύτερον, πρέπει οι επόπτε να έχουν την απαραίτητη ευελιξία στην εργαλειοθήκη του έτσι ώστε να είναι αποδοτικοί και να αντιμετωπίσουν και του ιδιοσυγκρασίε κριτικούς κινδύνους των ε, διαφόρων ε, ταμείων. Επίσης θα πρέπει στις προτάσεις μας για το δεύτερο σκέλος να ενισχύσουμε την εποπτική σύγκληση και να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στα βασικά σημεία σε επίπεδο εποπτικής δράσης. Τρίτον, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την κατάλληλη αρμόνιση κάποιων βασικών εποπτικών εργαλείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της μείωσης των κεφαλαίων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους οι οποίοι δεν καλύπτονται από τα λογιστικά τους λογιστικού κανόνε και αυτό κυρίω για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω. Τέταρτον, η πρόταση δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για την επόμενη εναρμόνιση του προληπτικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη πρόοδο στην εναρμόνιση τη διακριτική ευχαίρεια και των εθνικών εναλλακτικών σενάριων που προσφέρονται στα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε πω το Κοινοβούλιο εδώ θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θα μα βοηθήσει στην προσπάθεια τη διαπραγματεύση. Πέμπτον, απλούστευση κάποιων κανόνων για τις αμοιβέ, για την αποκάλυψη και θα πρέπει οι επόπτες να έχουν μια ευελιξία και διακριτική ευχέρεια με αναλογικότητα να εφαρμόσουν τους κανονισμούς. Θα πρέπει να διατηρήσουμε το ε, τους ίδιους κανόνες για όλους, το single rule book και είναι καλύτερο να μην, χρησιμοποιήσουμε, να μην τη δυνατότητα αυτή για να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μικρές τράπεζες. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς τι είναι μικρό, μικρή τράπεζα. Και επίση μια μικρή τράπεζα μπορεί να έχει υψηλού κινδύνου για του καταθέτε που δεν προστατεύονται. Και νομίζω ότι όπω είδαμε και με τι ισπανικέ τράπεζε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη χρηματοπιστική κρίση. Δεύτερον, για τι εξαιρέσει και τι απαιτήσει κεφαλαίου μέσα σε τραπεζικού ομίλου που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασυνοριακά. Αυτό θα μα επιτρέψει μια καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε πω η Τραπεζική Ένωση επιτρέπει αυτέ αυτές οι εξαιρέσεις να ε, προσφέρονται μέσα από τον SSM χωρίς να δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Λοιπόν, καταρχήν, θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε ως συμπέρασμα να ελαφρύνουμε τους υφιστάμενους κινδύνους και να ενισχύσουμε ε, τη σταθερότητα της τραπεζικής, ε, του τραπεζικού συστήματος στον, ε, στο χώρο του ευρώ. Θέλουμε συνεργασία στενή με υποπτικές και κανονιστικές αρμόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν αρκετές τράπεζες οι οποίες ακόμα χρειάζεται να κάνουν γρήγορα και αποφασιστικά βήματα έτσι ώστε τα στοιχεία ενεργητικού να ενισχυθούν και να είναι αξιόπιστα επιχειρηματικά μοντέλα και να μπορούν σήμερα να είναι αποδοτικέ στο σημερινό επενδυτικό περιβάλλον. Δεύτερον, οι νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εθνικό επίπεδο θα πρέπει να κάνουν βήματα εναρμονισμένα με τα σωστά εργαλεία έτσι ώστε οι επόπτε να έχουν την κατάλληλη ευελιξία έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν γρήγορα όπου είναι απαραίτητο. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. The first speaker is Brian. Ευχαριστώ. Πρώτος ο κύριος Μπράιν Χέις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήλθατε και πάλι στην Επιτροπή Οίκων. Σα ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Έπειτα από τα σχόλια του Προέδρου σχετικά με την επιτυχία της πρώτης εκαθάρισης της Banco Popular και όπως είπε ορθώς υπήρξε ιδιώτης αγοραστής και στέφθηκε η διαδικασία με επιτυχία βεβαίως. Γνωρίζετε όμως ότι το πρόσφατο τραπεζικό πακέτο ζητά αναθεώρηση της ε, υπάρχουσας εργαλειοθήκης για την εποπτεία όσον αφορά την εξυγίαση και την εκαθάριση και θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια όσον αφορά αυτή την πιθανή αναθεώρηση το, της εργαλειοθήκης για τα stress test ε, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας. Δεύτερον, τι θα πρέπει να κάνουν οι υπόπτες όσον αφορά την απόφασή τους για αυτήν την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, ιδίω ως προς το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί. Και ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω. Αναφερθήκατε στο ζήτημα του, των NPL, με τα κόκκινα δάνεια. Ε, στην Ιρλανδία το, το ποσοστό εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό ε, υπάρχει όμως μια ανησυχία στην Ιρλανδία και αλλού ότι δεν είναι όλα τα κόκκινα δάνεια το ίδιο. Ότι ε, δεν είναι όλα ε, δυνάμενα να, ε, να τύχουν αναδιάρθρωσης ή διαχείρισης. Το ερώτημα που ανακύπτει λοιπόν είναι, ο SSM θεωρεί, εξετάζει ότι υπάρχουν διάφορα, διάφορες κατηγορίες, διάφοροι τύποι μη εξυπηρετούμενων δανείων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα, εκείνα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που μπορούν να τύχουν διαχείρισης ε, θα έπρεπε να λάβουν και περισσότερο χρόνο. Αυτά ε, και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή της και, και τις δυσκολίες που περιγράψατε ότι αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Να μιλήσω πρώτα για το Banco Popular, γιατί μου δίνει τη ευκαιρία να απαντήσω και σε ορισμένα θέματα που ανέφερε ο Πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι δεσμεύομαι από όρους εμπιστευτικότητα σχετικά με τους κανόνες των ε, ισπανικών αρχών αλλά και βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Οπότε θα απαντήσω όσον αφορά τη διαδικασία του τι κάνουμε σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Πράγματι, λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση. Γι' αυτό και οικοδομήθηκε η Τραπεζική Ένωση, προκειμένου να μπορούν να επιλύονται προβλήματα έγκαιρα και να εξασφαλίζεται ότι αντιμετωπίζονται ε, με βάση το εκάστοτε κατάλληλο επίπεδο, θεσμικό επίπεδο. Είναι πολύ ευκολότερο φυσικά να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση όταν υπάρχει αγοραστή ή και αγοραστέ, υπάρχει και ανταγωνισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει έναν χρειαζόμαστε και η λύση είναι ότι το πρόβλημα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί αρκετά έγκαιρα. Γιατί αν χάσουμε χρόνο, ε, μπορεί η εκάστοτε τράπεζα, η υποεκαθάριση τράπεζα να μην ενδιαφέρει ε, τα, να μην ενδιαφέρει του αγοραστέ. τα, τα χαρτοφυλάκια τη δηλαδή, τα περιουσιακά τη στοιχεία. Όσον αφορά την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση που αναφέρατε, να σας πω ότι πρόκειται κάτι που προβλέπεται στην BRRD, αλλά δεν είμαστε εμεί επικεφαλεί αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, η ίδια η τράπεζα πρέπει να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να ε, διαθέσουν δημόσια χρήματα στην τράπεζα. Αν συμφωνήσουν οι δημόσιες αρχές, οι εθνικές αρχές, τότε ο Υπουργός Οικονομικών, γενικά το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας, θα ζητήσει από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και γνωρίζετε ποιοι είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις. Δημόσια, ένας σημαντικός όρος είναι ε, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημόσια χρήματα για να καλυφθούν οι απώλειες της, ε, της τράπεζας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταστεί βιώσιμη, μακροπρόθεσμα και να αντιμετωπιστούν ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και σε μια τέτοια διαδικασία ο SSM απαντά σε δύο μόνο ε, ερωτήματα. Αν δηλαδή η τράπεζα είναι φερέγγια, πρέπει να ανακηρυχθεί ως φερέγγια η τράπεζα. Ε, πρόκειται βεβαίως για μια απόφαση ε, στο χρόνο, την, κατά το χρόνο λήψης της ε, έχει σημασία το τι θα πούμε, όμως κοιτάμε και μακρόπνοα πώς μπορεί να εξελιχθεί μια τράπεζα. Και δεύτερον, πρέπει να καλύψουμε ε, τις ε, ε, ε επάρκειες, την, την επάρκεια που ενδεχομένως να χρειαστεί στη διαδικασία της εξυγίασης. Αυτό, αυτό κάνουμε, το λιγότερο το περισσότερο. Πάντως συνεργαζόμαστε με όλες τις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να στεφτεί η διαδικασία αυτή με επιτυχία, διότι κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμο ζήτημα. Όταν υπάρχει προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και όταν δαπανώνται ε, δημόσια χρήματα για να καταστεί μια τράπεζα βιώσιμη, φυσικά η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι επιτυχής ε, μεσοπρόθεσμα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως εναπόκειται ε, στην Κομισιόν να ελέγξει αν πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια. Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προφανώς δεν είναι όλα τα κόκκινα δάνεια το ίδιο το αντίθετο. Κάθε μη εξυπηρετούμενο δάνειο έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις ε, στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι συστηματικά κάνουν αυτό. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν ε, μεμονωμένοι πολίτες, ε, δανειοδοτούμενοι, άλλοι έχουν ενυπόθηκα δάνεια, ε, άλλοι χρησιμοποιούν διάφορα χρηματοδοτικά ή χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Υπάρχουν διάφορα είδη και τύποι δανείων, στις οποίες πρέπει να δοθούν διαφορετικές απαντήσεις, διαφορετικές λύσεις. Αλλιώς ε, αντιμετωπίζεται ε, κάθε υπόθεση, ιδίως αυτά τα χαρτοφυλάκια του παρελθόντος που, που κουβαλάνε δηλαδή αυτές τις δυσκολίες εδώ και πολλά χρόνια μαζί τους. Φυσικά θα χρειαστεί χρόνο. Αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι οι τράπεζε θα κινηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φυσικά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ. Εκτό από φιλόδοξοι, πρέπει να έχουμε κατά νου και κάτι το οποίο να είναι και εφικτό. Ε, γι' αυτό και εξετάζουμε τις, ε, ε τις στρατηγικές και τα σχέδια που μας παρουσιάζουν οι τράπεζες. Κάποιες φορές είναι πιστικά, κάποιες φορές όχι τόσο και όταν δεν είναι πιστικά τα σχέδια που μας υποβάλλουν οι τράπεζες, ε, τις καλούμε να ξανακάνουν την, ε, τη δουλειά από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη ερώτηση εγώ. Και συνεχίζω. Στην υπόθεση του Banco Popular. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι δεν μπορείτε να πείτε πολλά σε μια δημόσια συνεδρίαση αλλά έχει νόημα να προχωρήσουμε εις βάθος το διάλογο αυτόν. Και έτσι ξεκινώ. Ο μηχανισμός σταθερότητας είχε γνώση των προβλημάτων της τράπεζας και αν ναι, είχαν γίνει αυτοψίες είχαν γίνει αυτοψίες εάν έγιναν από επόπτες που δεν ανήκαν στην ίδια εθνικότητα αλλά από ομάδες απαρτιζόμενες από επόπτες διαφορετικών ε, εθνικοτήτων έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας πιο ευνοϊκής μεταχείρισης και εάν έγιναν όλα αυτά γιατί θεωρείτε ότι απέτυχε το σύστημα να εντοπίσει Προβλήματα τα οποία άλλωστε χωρίς να υπάρξει πίεση εμφανίστηκαν. Επίσης, είπατε ότι θα έπρεπε να έχετε περισσότερες εξουσίες ως προς την ε, παρέμβαση προληπτικά στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Πάντως έχετε αρκετές εξουσίες και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η διαδικασία η διαδικασία που είχατε στη θέση σας υλοποιήθηκε. Τότε γιατί δεν λάβατε κάποιο μέτρο για αντιμετωπίσετε στο πλαίσιο των ήδη φυσταμένων εξουσιών σας των προβλημάτων. Γιατί δεν έγιναν περισσότερα από όσα έγιναν. Εάν είχε η τράπεζα πρόβλημα και το γνωρίζατε, γιατί δεν δράσατε και δεν αντιδράσατε ως ε, χρειαζόταν ή γιατί δεν το γνωρίζατε. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό σημείο καμπή αυτή η υπόθεση, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία βεβαίω που δεν έχει ολοκληρωθεί. Τραπεζική Ένωση, Μπάξη, Έντις, Ντέμρελ, δεν τα έχουμε όλα αυτά. Είμαστε μόνο σε μια ε, πρόβλεψη πρόορης παρέμβασης. Ε, μήπως όμως θα έπρεπε να καταλήξουμε συμπεράσμα ότι αν κάτι δεν έχει λειτουργήσει καλά Ομολογούμε ότι αυτό οφείλεται σε κάποια ελλείμματα, ανεπάρκεια και αν φτάσουμε σε αυτό, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα και την ανεπάρκεια. Ευχαριστώ πολύ σε σχέση με τις ερωτήσεις τις σχετικές με την Banco Popular. Ε, τονίζω για άλλη μια φορά ότι έχω ε, περιορισμούς λόγω της ε, του απόλυτου χαρακτήρα όλων αυτών. Βεβαίως και γνωρίζαμε ήδη από το stress test, από το τεστ αντοχής του 2016 της ΕΜΠΑ, της ΕΤΑ δηλαδή Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, είχε φανεί στο, η ανάπτυξη κεφαλαίου, κεφαλαίου ήταν ε, επίσης σημαντική, με 600 σημεία σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων. Άρα γνωρίζαμε και παρακολουθούσαμε την υπόθεση αυτή στην περίοδο της εποπτείας μας. Επίσης θα θυμάστε ίσως ότι τα τεστ δοκιμής δεν ήταν ε, ασπρομαύρο ή πέρασε κόπικες το 2015-2016. Η ανάπτυξη πάντως κεφαλαίου ήταν ε, ήδη ορατή. Η διασπορά κεφαλαίου καλύτερα. Και πάλι αν δεν κάνω λάθος, είχε αρκετά καλά αποτελέσματα. Πέντε δις πρόσθετου κεφαλαίου είχε μπορέσει να ε, αναπτύξει η τράπεζα. Αρκετά δηλαδή έως και σημαντικά ποσά. Επίσης, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των σενάριων για τα τεστ αντοχής. Ε, ο μηχανισμός έχει δικαίωμα ψήφου στην ΕΤΑ. Και η ΕΤΑ δεν είναι το μόνο όργανο το οποίο συμφώνησε στην ε, διαπίστωση αρνητικού σεναρίου. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να έχουν τα εποπτικά συμβούλια σύγκρουση συμφερόντων. Γι' αυτό και είναι καλό που δεν έχουν γνώμη στην υπόθεση αυτοί δεν ε, ψηφίζουν. Αλλά στην υπόθεση της νομοθεσίας Λιοβιέρη που είναι βέβαια η βάση αυτής της ε, κρίσης, η κρίση στην Ισπανία δεν ε, προέκυψε λόγω της ενίσχυσης της φούσκας. Ήταν ήδη ένα σύστημα σε ανάπτυξη και μάλιστα κατασπάραξε πολλές τράπεζες. Επομένως, ε, ήταν πιθανόν, ήταν δυνατόν να πιθανολογηθεί ότι ένα αρνητικό σενάριο για την Ισπανία θα μπορούσε να υλοποιηθεί γιατί η πραγματική ζωή είναι πάντα πιο σκληρή από ένα τεστ αντοχής όσο σκληρό και είναι αυτό. Όπως είπατε όμως πρόεδρε, κάναμε πολλά κι εμείς με τις αυτοψίες μας. και νομίζω ότι αυτό είναι ορατό. Υπάρχουν ε, σχετικές ε, δημόσια διαθέσιμες λογοδοσίες, εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, σε σχέση με την ε, δραστηριότητα της εποπτείας της τραπεζικής. Όπως είπατε και εσείς, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να είχαμε μπορέσει να εντοπίσουμε πού ήταν το δικό μας φάλμα αλλά δυστυχώς δεν είμαι σε θέση, έστω και έχοντας ε, αφήσει αυτή την υπόθεση στο παρελθόν και γνωρίζοντας ε, και μπορώντα να εξετάσω τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά, δεν μπορώ να το πείσω το δικό μας λάθος. Και είναι η πρώτη φορά μέσα σε τρία και περισσότερα χρόνια που ε, κηρύσσεται αφαιρέγγια μία τράπεζα. Ναι, αλλά είναι μόνο μία. Και επιπλέον θα ήθελα να πω για φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ποτέ δεν μπορούσε να κηρυχθεί αφαιρέγγια ή πιθανώς αφαιρέγγια μια τράπεζα. Τα εργαλεία που έχουμε στη θέση μας για αυτόν τον λόγο έχουν σχεδιαστεί, γιατί υπάρχουν φορές που πρέπει μια τράπεζα να εξαλειφθεί, να εξαφανιστεί, γιατί το Συμβούλιο του Διοικητικό δεν έχει λάβει τις αποφάσεις που οφείλει να λάβει. Σημαντικό πάντως είναι να υπάρχει ε, το πλαίσιο η τράπεζα, το Συμβούλιο Εποπτείας, ο μηχανισμός, να υπάρχουν όλα αυτά που θα λειτουργούν κατά τρόπο απρόσκοπτο θα επιτρέπουν την συνέχιση της λειτουργίας της τράπεζας, η οποία, ξέρετε, την επόμενη μέρα ξανά τις πόρτες της και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, χωρίς να απορροφήσει δημόσιο χρήμα, χωρίς να προξενήσει κλειδονισμούς. Και με όλη την ε, με τριοφροσύνη, γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να το πει κανείς αυτό, πρέπει να πω ότι εμείς τουλάχιστον τη δοκιμασία του πλαισίου στη συγκεκριμένη κατηγορία μια σκληρής, δύσκολης, πόδινης απόφασης την περάσαμε. Με επιτυχία. Ο πρόεδρος, ε, με λίπο μου θα πω ότι δεν συμφωνώ μαζί σας και θα ήταν καλύτερο μηχανισμός να αναγνωρίσει στα σχόλια του τα προβλήματα να τα εντοπίσει, να προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση. Παρακαλώ εσείς. Μια ερώτηση, Πρόεδρε, κύριος Φεκμάκ. Είπατε ότι δεν έχουμε το MRL. MRL. Υπάρχει νομοθεσία, λέει ο κύριος Γουαλτιέρη, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως στις τράπεζες, γιατί όπως ξέρεις, μα το έχουμε το MRL, μα βεβαίως επί χάρτου, βεβαίως και υπάρχει. Μα οι κανόνες υφίστανται. Επειδή είπατε ότι δεν, έχει, δεν υπάρχει μερέλ. Να, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα περάσει χρόνος μέχρι να αναπτύξει πλήρη λειτουργία αυτή η νομοθεσία. Και εάν ήταν να κηρύξει πάυση πληρωμών η τράπεζα αυτή, θα έπρεπε να χτυπήσει τις καταθέσεις. Να χτυπηθούν μάλλον οι καταθέσεις ναι, αλλά την έχουμε, μάλιστα. Κύριος Λούλτς. Θα συμφωνήσω με τα όσα είπατε, Πρόεδρε, σε μεγάλο βαθμό και θα ήθελα να καλωσορίσω και την κυρία Νουή. Τώρα, για τον Banco Popular θέλω να πω δύο λόγια ακόμα. Πριν από δέκα μέρες διάβασα μία ανακοίνωση της Αντιπροεδρίας της ΕΚΤ και εκεί δήλωσε ο λόγος που οδήγησε στην απόφαση αυτή είχε να κάνει ε, με ε, το, τη μείωση των ποσών καταθέσεων και ήταν η ρευστότητα η οποία μας οδήγησε σε τούτη την απόφαση. Και γι' αυτό θεωρούμε πως είναι πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε στο σημείο αυτό και να δούμε αν η έλλειψη ρευστότητα μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος ενδεχόμενης χρεοκοπίας ή ε, κινδύνου χρεοκοπίας για μια τράπεζα. Ίσως λοιπόν υπάρχουν κάποια στοιχεία, επειδή όλα αυτά γίνονται στην Ισπανία, τα οποία, δεν, τα οποία μου έχουν διαφύγει, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια μέτρα και ποια κατόφλια λάβατε υπόψη για να καταλήξετε στην απόφαση αυτή. Και κυρίως γιατί έχουμε ακόμα κάποιες τέτοιε περιπτώσεις στην Ευρωζώνη, σε εκκρεμότητα και σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί θα ήθελα να συγκρίνω με την μειούμενη ρευστότητα που διαπιστώνουμε σήμερα σε τρεις Ιταλικές τράπεζες. Μοντεπάσκι, Banco Popular de Vincenza, ε, τράπεζες οι οποίες ε, οι επενδυτές και οι καταθέτες αντιμετωπίζουν με νευρικότητα, οπότε τι κάνει κανείς για τις τρεις αυτές Ιταλικές τράπεζες, εάν λάβει κανείς και ακολουθήσει την ίδια λογική ε, με τα κατόφλια ρευστότητα και τα λοιπά που είχατε με τον Banco Popular. Ή διαφέρουν αυτέ οι τράπεζε από τον Banco Popular και με ποιο τρόπο τότε. Αυτή νομίζω είναι και η πιο σχετική ερώτηση. Ναι, γιατί δεν πέρασαν καταρχήν από τα stress test οι τράπεζες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς Συχνά όταν αυτή τη στιγμή, σε κάποια στιγμή κινδυνεύει μια τράπεζα, η ρευστότητα είναι και το τελευταίο, το τελευταίο σύμπτωμα της ασθένειας. Ε, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο σωματοποιείται η ασθένεια. Δεν είναι μόνο όμως θέμα ρευστότητας, αυτό είπα και προηγουμένως. τα δύο τελευταία τρία χρόνια είχαν επιπλέον δις κεφαλαίων, είχαν γίνει δηλαδή ενέσεις πέντε δις ε, σε όλη αυτή την περίοδο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ρευστότητα. Εάν λοιπόν η τράπεζα αυτή είχε πολιθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο, Με συγχωρείτε, η πώληση λοιπόν και η απόφαση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο είχε να κάνει περισσότερο με κάποιες δομικές αποφάσεις παρά από αυτό το τελευταίο βήμα που επαναλαμβάνω ήταν και το τελευταίο σύμπτωμα μιας βαθιάς ασθένειας. Τώρα, κατόφλι. Υπάρχει κατόφλι ρευστότητας. Νομίζω πως ουσιαστικά το τελευταίο που πρέπει να αποφύγουμε είναι κάποια στιγμή η τράπεζα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τα δικά της δάνεια. Και όλα γίνονται βέβαια ε, ηλεκτρονικά πια, αλλά να το πω έτσι, να μην κατεβάσει ε, τα ρολά. Το τι θα γίνει με τις τράπεζες που αναφέρατε εσείς, ε, και πότε εμείς θα άρουμε ε, την, ε, την δυνατότητα λειτουργίας και το τι γίνεται με τα στοιχεία ενεργητικού μιας τράπεζας που κινδυνεύει, όλα αυτά γίνονται σε περιπτώσεις που κάποια τραπεζικά καταστήματα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους κτλ. Αυτός είναι ο ορισμός ε, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ε, στο νομικό πλαίσιο για την προληπτική επικοινωνιοποίηση. Τώρα, για μια τράπεζα, όσο μπορεί να εξυπηρετεί τι δικέ τη υποχρεώσει, δεν μπορεί να θεωρηθεί κανεί πω κινδυνεύει. Αν δεν μπορεί όμω να τι αντιμετωπίσει ή αν θεωρούμε πω το άμεσο μέλλον δεν μπορεί, τότε ναι. Τότε θεωρείται ότι ενδέχεται να κινδυνεύει. Και όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσει να σα πω πω το περιθώριο λίγο μόνο που έχουμε δεν είναι μεγάλο. Σε τέτοιε περιπτώσει, δυστυχώ πρέπει να αναλάβουμε δράση. Καλύτερα βέβαια αυτό να γίνει Σαββατοκύριακο, ιδίω σε χώρε όπου δεν υπάρχει μορατόριο, έτσι ώστε ε, να δούμε πώς θα εξυπηρετηθούν και με ποια σειρά οι καταθέτες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και με τον Banco Popular χρειάζεται και να λάβουμε μία απόφαση. Ευχαριστώ πολύ, ο Ραμόν Τρεμόσα. Καλώς ορίσατε, κυρία Νουή, στο Κοινοβούλιο, μια φορά ακόμα. Ε, Έχω δύο ερωτήσει σχετικά με, τον, με την Banco Popular και να απαντήσω και στην συνάδελφα των. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στην Ισπανία ε, δημόσια χρήματα για καθάριση ε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης έδρασε γρήγορα. Το χαιρετίζουμε. Τον, ε, τον, την επόμενη χρονιά η τράπεζα Σανταντέρ θα ε, ε, της επιτραπεί να πληρώσει λιγότερους φόρους προκειμένου να ε, ε διευκολυνθεί. Ωστόσο, όπως είπε ε, ο πρόεδρος, ε, ε, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν ήταν ζήτημα φεργιότητας αλλά ζήτημα ρευστότητας. Υπήρξε μαζική εγκροή κεφαλαίων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, θα διερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες που εμφανίστηκαν στον τύπο την προηγούμενη ε, εβδομάδα. Ο Υπουργό Γκίντο είπε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν περιφερειακές κυβερνήσει, ακόμη και το ασφαλιστικό σύστημα τη Ισπανία, που ε, προκάλεσε αυτή τη μαζική εκροή κεφαλαίων. Δεν υπήρχε τίποτα στους δρόμους, στα ATM, δεν υπήρχαν μικροί καταθέτες, δηλαδή αποταμιευτές οι οποίοι πήγαιναν στα υποκαταστήματα για να πάρουν τα χρήματά τους. Αντιθέτως, φαίνεται ότι κάποιες περιφερειακές, τοπικές κυβερνήσεις, δημοτικές ε, περιφερειακές αρχές, ήταν εκείνες οι οποίες απέσυραν δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια δύο μέρες πριν από την παρέμβαση. Σας ρωτώ λοιπόν, θα διερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες. Την ε, πιθανή δηλαδή ε, απόφαση που προκάλεσε την κρίση ρευστότητα της Banco Popular. Και δεύτερον, με το ε, μη εξυπηρετούμενο δάνειο της, ε, της ε, Banco Popular και με δεδομένα όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτή η εξηγένση που κάνατε θα αποτελέσει μοντέλο και για το μέλλον και αν ναι, για ποιο λόγο θα, θα ε, κληθεί κανείς να επενδύσει ποτέ ξανά σε τέτοιου είδους τράπεζες όπως η Banco Popular με τόσο μεγάλο μη εξυπηρετούμενα ε, δάνεια. Για το πρώτο ερώτημα, Υπήρξαν κάποιοι πιο ισχυροί ε, καταθέτες οι οποίοι πράγματι απέσυραν ε, τις καταθέσεις τους ε, όπως λέτε εσείς δηλαδή εγώ δεν είμαι αστυνομικό, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω προφανώς η ισπανική δικαιοσύνη και οι αρχές εποπτείας αγοράς της Ισπανίας θα πρέπει να διαρευνήσουν αυτού του είδους τις και να λάβουν μέτρα αν κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Όσον αφορά τα κόκο και το, τα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτές ακριβώς είναι οι, οι, ανησυχίες που θα κληθούν τα εργαλεία μας, όπως το MRL, να αντιμετωπίσουν. Έχουν υψηλές αποδόσεις, όπως ε, τα ε, τα ομόλογα για παράδειγμα, φυσικά πρέπει κάθε αγοραστής τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικού εμ, προϊόντος να γνωρίζει. Δεν θα πρέπει όμως κάθε ε, λιανοπολιτής να μπορεί να τα αγοράζει και να τα πωλεί έτσι με, με μεγάλη ευκολία αυτά τα προϊόντα, διότι ε, εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα. Χρειάζεται να εξασφαλίζεται μια μεγάλη διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών και των καταθετών. Αλλά αυτά είναι πάντοτε ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε στις τράπεζες όταν αυτές πλησιάζουν στην εξυγίασή τους. Θα πρέπει ωστόσο οι πολίτες, οι αγοραστές να, είναι, ε, να έχουν πλήρη επίγνωση αυτών των περιστάσεων όταν αγοράζουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Κάτι ακόμη. Σας ρώτησα αν ο SSM θα διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις της, απο... της απόφασης της Ισπανικής κυβέρνησης. Μου απαντήσατε όχι. Δεν γνωρίζω. Διότι, ναι, μπορεί να ήταν οι περιφερειακές απαντήσεις, μπορεί να ήταν ασφαλιστικά ταμεία. Όχι, ναι, κυρία Νούη, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Άλλες αρχές, όπως οι αρχές αποκτήρια αγοράς της Ισπανίας ή η Ισπανική δικαιοσύνη, ε, καλούνται να διερευνήσουν. Είπατε όμως πριν από τρεις εβδομάδες ότι η Banco Popular ήταν ε, φερέγγια και το αποσύρατε αυτό πριν από δύο εβδομάδες. Πότε ακριβώς συνέβη αυτή η αλλαγή ε, και πώς ακριβώς θα διερευνηθούν ε, αυτές οι καταγγελίες. Ξανααπαντώ ότι είναι οι αρχές εποπτήσεις αγοράς που πρέπει να, δώσουν, να κάνουν τη διερεύνηση. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Η δική μας ε, άποψη είναι πως η λύση που έδωσε που δώσαμε για το Banco Popular δημιουργεί πολλές αμφιβολίες και για την κυβέρνησή μας και για την ΕΚΤ και για την Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας και αυτός ο πολύ θριαμβευτικός τόνος πραγματικά δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητός γιατί και η διαδικασία είναι περίεργο. Το βράδυ πριν αποφασιστεί η λύση αυτή έγιναν μεγάλες κινήσεις καταθέσεων που αποδεικνύει πως κάποιοι είχαν πληροφορίες ε, εσωτερικές ε, και ήταν οι μικρομέτοχοι οι οποίοι έχασαν πρώτοι. Γιατί αν μιλά κανεί για το ποιον έχασε, θα πρέπει καταρχήν να μιλήσουμε για όσου δούλευαν στην τράπεζα αυτή, οι οποίοι ενδεχομένω θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση προσωπικού. Και αν δεν έφτανε αυτό, θα έπρεπε να δούμε πώς για μια φορά ακόμα αυτή, η, αυτός ο λογιστικός έλεγχος που ήδη καταδικάστηκε για το πώς επόπτευε την Μπάνκια και πάλι και πάλι επέτρεψε αυτού του είδους τις συναλλαγές παρουσιάζοντας μια έκθεση που επιτρέπει για ένα ευρώ να πολιθεί ε, η Μπάνκο Σανταντέρ που στη δική μας χώρα θεωρήθηκε ε, απαράδεκτο. Μα, συγγνώμη, είχαν γίνει stress τεστ με το Banco Popular και είχε βγει λάδι. Και νομίζω ότι ο συνάδελφος το είπε, ο υπουργό ε, Οικονομικών είπε, είναι μια υγιής τράπεζα. Λοιπόν, εάν πρόκειται ε, να, α, να θεωρήσετε εσείς τα stress τεστ, να μας το πείτε, γιατί δεν μοιάζουν να πετυχαίνουν. Επίσης, η λύση για τον Banco Popular ανοίγει το δρόμο για αγωγές, μια και δεν έγινε... Ε, δεν έγινε σεβαστή η αρχή το ότι η λύση δεν θα πρέπει να είναι χειρότερη από οποιαδήποτε αποτέλεσμα ε, δικαστικής προσφυγής. Και τι γίνεται με τη συγκέντρωση στο χρηματοπιστωτικό τομέα στη χώρα μου. Δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο κάτι τέτοιο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβολικά μεγάλες τράπεζες που είναι τόσο μεγάλες που είναι αδύνατο να τις αφήσουμε να χρεοκοπήσουν. Κάτι το οποίο έχουμε δει στο παρελθόν και το οποίο αυξάνει το συστημικό κίνδυνο. Θεωρείτε εσείς πως η απορρόφηση αυτών των μεσαίων τραπεζών από τις μεγάλες τράπεζες είναι θετική συνέπεια αυτού του ενιαίου συστήματος ε, αντιμετώπισης. Υπάρχει δηλαδή συστημικός κίνδυνος από, αυτά, από αυτές τις υπερβολικά μεγάλες τράπεζες. Ελπίζω να σας κατάλαβα γιατί μιλούσατε πολύ γρήγορα και νομίζω ότι αποτελέσατε και πρόκληση για τους γερμηνείς. Λοιπόν, τα όσα είπατε για την κίνηση, μεγάλη ε, με κινήσεις καταθέσεων το προηγούμενο βράδυ, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό. Σίγουρα υπάρχουν ε, περιθώρια για την ισπανική δικαιοσύνη να κινηθεί και να ερευνήσει κατά πόσο είχαμε τέτοιου είδους κίνηση καταθέσεων λόγω ε, εσωτερικής πληροφόρησης και νομίζω ότι καλό θα ήταν η μικροκαταθέτες δεν είναι σε άσχημη θέση γιατί κανείς καταθέτης αυτή τη στιγμή δεν, έλα, δεν έχασε ούτε ένα σέντ. Όλοι προστατεύτηκαν. Εκτός βέβαια αν οι μικροκαταθέτες ή οι, οι μικροκαταθέτες είχαν στα χέρια τους, ήταν και μικρομέτοχοι παράλληλα. Αλλά ξέρετε ότι αυτό δεν είναι τόσο ασφαλές, το να έχει κανείς ε, μετοχές... Ε, ε, όταν κάποια τράπεζα κινδυνεύει είναι ιονή επικίνδυνο. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα διδάγματα ε, και το λέω αυτό προς υπενθύμηση. Για τις αγωγές, ναι, είμαι σίγουρη πως θα έχουμε πάρα πολλές. Και ας αφήσουμε το μέλλον να αποφασίσει, να δούμε αν θα είναι ε, κάποιος, κάποιοι, ένας θεσμός, ε, που θα αποταθούν στην δικαιοσύνη και η οποία κατόπιν θα αποφανθεί. Για την συγκέντρωση και το κατά πόσο είναι υπερβολικά μεγάλες για να τις αφήσουμε να χρεοκοπήσουν, μπορεί. Για μένα όμως δεν έχει να κάνει με το μέγεθος, αλλά έχει να κάνει με, την, με το πόσο περίπλοκες είναι οι μεγάλες τράπεζες, πολύ πιο περίπλοκα, περίπλοκες οντότητες από τις μικρές, πιο εξελιγμένες, πιο εξωτικές τραπεζικές επιχειρήσεις, χρηματιστηριακής επιχειρήσεις, πολλά στοιχεία εκτός ισολογισμού και συναλλαγές εκεί. Λιγότερη διαφάνεια είναι συναλλαγές οι οποίες όντως μπορεί να δημιουργούν κινδύνους. Εδώ μιλούμε όμως για τέτοιου είδους ε, τράπεζες, γιατί αν μιλήσουμε για τη Σανταντέρ και για τις άλλες στις οποίες αναφερθήκατε, Εντάξει, αν οι τράπεζες αυτές δανείζουν ε, ε, με εγγυήσει ε, ακίνητα, υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι περισσότερες οι προκλήσεις εδώ, τουλάχιστον σε επίπεδα υποπτίας. Οπότε στην περίπτωση αυτή, όχι, δεν ανησυχώ έτσι όπως προτείνατε. Συγγνώμη, δεν έχουμε όλο Thank Ευχαριστώ, κύριο Σούρτασον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε εδώ, κυρία Νουή. Σήμερα ε, έχω τι εξή ερωτήσει. Νωρίτερα, όταν αναφερθήκατε στην οντότητα παρέμβαση για το άρθρο 13 του κανονισμού του SRM, δηλώνει ότι θα πρέπει να ενημερώσετε την SRB όταν υπάρχει μια ε, προηγούμενη παρέμβαση και με τους όρους του άρθρου 27 όπου ρητά αναφέρεται το όταν υπάρχει ταχεία επιδείνωση της ε, χρηματοοικονομικής κατάστασης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος περιλαμβανομένων και των προβλημάτων ρευστότητα, μία πρόορη παρέμβαση είναι απαραίτητο εργαλείο. Ερωτώ λοιπόν υπήρξε ε, πρόορη παρέμβαση από τον SSM στην περίπτωση του Banco Popular, ναι ή ου και αν ναι πότε, εάν ου, για ποιους λόγους δεν έλαβε χώρα αυτή η παρέμβαση, αφού ορίζεται στους κανόνες. Επίσης, τα προβλήματα ρευστότητας της τράπεζας. Υπήρξε στιγμή όπου η Banco Popular είχε ποσοστό ρευστότητας πολύ χαμηλότερο από το υποχρεωτικό όριο. Ερωτώ λοιπόν, από ποια χρονική στιγμή η Banco Popular εξεδήλωσε αυτό το χαμηλότερο από το υποχρεωτικό επίπεδο ποσοστό ρευστότητας και με βεβαίω ότι έχετε σχετική ενημέρωση γιατί αφού έχει την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ισπανική Τράπεζα την ΕΛΑ ή η Banco Popular πρέπει να είστε εν γνώση. Πότε λοιπόν, ποιο είναι το χρονικό σημείο, διότι είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουμε από ποια στιγμή και μετά ε, λειτουργούσε με επίπεδο χαμηλότερο της υποχρεωτικής ρευστότητας η Banco Popular. Και επίσης το 2016 η κάλυψη αυτή ήταν, 1, ήταν 100 1,187%. Ήταν 187%. Πολύ περισσότερο δηλαδή από το απαιτούμενο. Άρα πότε έπεσε τόσο χαμηλά. Και επίσης σε σχέση με τη διαχείριση του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου. Καταστροφή. Και αποχώρησε μέλος του με 73 εκατομμύρια ευρώ σύνταξη. Έχει συγκλονιστεί όλη η Ισπανία. Και ιδιαίτερα οι μικροκαταθέτες των οποίων έχουν ε, ε, χαθεί οι αποταμιεύσεις. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μήπως θα έπρεπε και, αυτά τα, και αυτές οι αποδοχές να περνούν στη διαδικασία της αυτοδιάσωσης. Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα παρέμβασης υπάρχουν δύο κανονισμοί, CRD4-4 και BRD. CRD4-CRR και BRD. Λοιπόν, σε σχέση με το BRD η απάντησή μου θα είναι αρνητική. Γιατί, Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ε, ακολουθούμε την αρχή της αναλογικότητας στη δράση μας. Δηλαδή πρέπει να σταθμίσουμε Μάλλον πρέπει να αναλάβουμε την ελάχιστη απαιτούμενη δράση για να φτάσουμε στον επιδιωκόμενο σκοπό. Τα δε δύο καθεστώτα που οι τράπεζες τα βλέπουμε διαφορετικό, τα αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο, με το CRD4 έχουμε, και το CRR έχουμε ε, πρόωρα μέτρα ή πρόημα μέτρα παρέμβασης που θεωρούνται κάτι το τετριμένο, ενώ με το BRD οι τραπεζίτες θεωρούν ότι έχουν υποστεί βαρύ πλήγμα. Είναι δυνατόν όντως να αναπτυχθούν τα σχετικά μέτρα του BRD, αλλά για να σεβαστούμε την αρχή αυτή της αναλογικότητας με την ελάχιστη εποπτική δράση, απέστειλα εγώ επιστολή στον νομοθέτη την Επιτροπή για να εξηγήσω ότι η σύνταξη των μέτρων, η διατύπωση των μέτρων προώρης παρέμβασης για μένα αποτελεί σημαντικό πρόσκοπμα γιατί δεν είμαι σε θέση να εντοπίσω ευχερός τους όρους και τις προϋποθέσεις που τους οποίους μπορούν να, να ενεργοποιηθούν τα μέτρα. Και πολλοί από τα μέλη του Συμβουλίου μας ε, μένουν σε βεβαιότητα λόγω ακριβώ τη ασάφεια στη διατύπωση εάν είναι η στιγμή κατάλληλη για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα, πώ είναι πολύ νωρί, πώ είναι πολύ αργά. Και επίσης Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μπορούμε να ανοίξουμε τα βιβλία μας με το SRB και με την ε, Εθνική Αρχή Εποπτείας δηλαδή ε, πολύ πολύ νωρίτερα και σε σχέση με τα μέτρα παρέμβασης του BRD. Γιατί πάντα αυτή η συνεργασία είναι με, την, με βάση το αν έχουν κάποιο ένομο συμφέρον ή ε, λόγο να ενημερωθούν. Πρέπει λοιπόν με αυτό το γνώμονα να δρούμε. Εάν είναι εύλογο να ενημερωθεί η αρχή εποπτείας. Και αυτό, όπως είπα, έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των πιο σκληρών μέτρων του BRD. Αντίθετα με το, με το CRD4, το CRR, δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις και ενδείξεις ότι μπορούμε, εάν δεν αλλάξουν πορεία, γιατί η πορεία που έχουμε επιλέξει είναι ε, εσφαλμένη, μπορούμε λοιπόν εμείς να τους ε, προωθήσουμε, να τους υποχρεώσουμε σε ε, εκαθάριση. Τώρα για τα επίπεδα του... η διακύμανση των καθημερινών επιπέδων ε, ρευστότητας, δεν μπορώ να σχολιάσω για λόγους απορρίτου, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχουμε τη δυνατότητα της ε, εκαθάρισης μπορεί αυτό να προχωρήσει με πιο γρήγορους ή πιο αργούς ρυθμούς κατά περίπτωση. Όταν είναι πιο γρήγοροι οι ρυθμοί, αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι έχουμε παρακολουθήσει ε, κατά πόδα στην κρίση, ενώ αντίστροφα, εάν ε, είναι πιο βραδύς οι ρυθμοί, μπορεί αυτό να οφείλεται στο ότι ήμασταν πιο επιφυλακτικοί ως προς την δράση αυτή. Και αν δούμε ότι δεν υπάρχει ε, κίνδυνος, μπορούμε να ε, αλλάξουμε συμπεριφορά. Μάρκο Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Στα Ιταλικά, αν έχετε την καλοσύνη να βάλετε τα ακουστικά σας. Στην ε, εισαγωγική σας παρέμφαση είπατε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να επιταχύνουμε του ρυθμού μα βεβαίω. και συμφωνώ ότι έχουμε να κάνουμε με σοβαρό πρόβλημα και εν προκειμένου έχουμε να κάνουμε με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αλλά όταν η κατάσταση έχει στρεβλωθεί τόσο από τις δύο τράπεζε, οι οποίε έχουν κατά κάποιο τρόπο απαλλαγή από το βάρο των ισολογισμών των προηγουμένων ετών, των δημοσίων χρεών και αυτό το λέω ιδιαίτερα και για τις ταλικές τράπεζες που έχουν ήδη σημαντικά σημαντικά ποσοστά μη εξυπηρετωμένων δανείων. Αλλά το να λέμε ότι θα πρέπει με πολύ ταχύς ρυθμούς να εκαθαριστούν, αυτό συνεπάγεται ότι ξεπουλούνται σε τιμές ε, πολύ χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία. Και αυτό συνεπάγεται με τη σειρά του μια συνθήκη κρίσεως και στρες, πίεσης δηλαδή τέτοια, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα και των ε, πιστοτικών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που μπορεί να είχαν ήδη μια κάποια δυσκολία να τα βγάζανε πέρα, αλλά ταυτόχρονα τώρα παίρνουν ένα πλήγμα τόσο βαρύ που δεν μπορούν παρά μόνο να βγουν σε καθάριση. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους πιέση μόνο επιτάχυνση της ε, εκαθάρισης ε, και, της, ε, και ενίσχυσης κατάστασης μπορεί να οδηγήσει. Επίσης, τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν και άλλα στοιχεία κινδύνου που είναι και δωδεκαπλάσια, συστημικός κίνδυνος δηλαδή για την ευρωπαϊκή οικονομία, δωδεκαπλάσιας αξίας από αυτήν των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω γιατί εξακολουθείτε να εστιάσετε την προσοχή σας μόνο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τους άξονες δεύτερου και τρίτου επίπεδου, που είναι πολύ μεγαλύτερη αξία τους. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όταν ε, είπατε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αναλάβει δράση νωρίτερα, ε, δεν καταλαβαίνω που, μπορεί να ήταν η πιο γρήγορη δράση μας. Το 2014 άρχισαμε να το εξετάζουμε, έφτασαμε στο 2017, έχοντας περάσει μέσα από μια μακρά διαδικασία, δημοσιοποίηση κατευθυντήριων γραμμών, διαβουλεύσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές, Ζητώντα από τι Τράπεζε γιατί τώρα σε αυτό το στάδιο είμαστε από τις τράπεζες, ε, τράπεζες να μα κοινοποιήσουν τα δικά τους ε, πλάνα, σχέδια για την αντιμετώπιση των ε, μη εξυπηρετουμένων δανείων και ε, θέλω να πω ότι ναι, όντως δεν μπορεί να κρατήσει επί δεκαετίες αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στην ταχύτητα που επιδιώκουμε. Άρα λοιπόν αξιολογείται η τράπεζα και αν η τράπεζα, όπως και κάθε μαθητής με σε μια τάξη, έτσι, μπορεί να μην είναι κανείς άριστος, αλλά αν τα πάει καλά και έχει υποβάλει ένα σχέδιο σχετικά λογικό, δεχόμαστε ότι έχει κάνει σωστές επιλογές. Επίσης μιλήσατε για τις τιμές ε, στην εκαφάριση, ότι δεν είναι αυτές που θα θέλανε οι τράπεζες. Μα ναι, είμαστε σε, βρισκόμαστε σε οικονομία αγοράς. Έχουμε πολιτεί όπως έχουμε και αγοραστεί. Και από αυτούς καθορίζεται τιμή. 900 εκατομμύρια μη εξυπηρετουμένων δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μειούμενη τάση βέβαια, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Ε, σημαίνει πως η ισχυρή διαπραγματευτική θέση έχει ο και όχι ο πολιτής της τράπεζας, η πολλουμένη τράπεζα. Και όντω είναι ε, απογοητευτικές οι τιμές. Και εμείς πολλές φορές αισθανόμαστε απογοήτευση. Γιατί βεβαίω όσο πιο πολλά χρήματα μπορέσουν να αποκομίσουν την πώληση του οι τράπεζε, τόσο πιο ισχυρέ θα είναι. Και αντιλαμβάνομαι βεβαίω ε, τα επιχειρηματά σα, αλλά ακριβώ αυτό θα συμβεί και σε σχέση με εκείνους που θα πουλήσουν πρώτοι, γιατί οι τελευταίοι θα έχουν μείνει και στα χαμηλότερα επίπεδα της ε, αγοράς. Για, τα επίπεδα, για τον ιδιωτικό επίπεδο 2 ή 3. Εγώ θα προτιμούσα να μην είχαν συνδεθεί τα δύο ζητήματα, γιατί είναι σαν να μου λέτε, ε, σε παρακαλώ, ε, κάνε τα στραβά μάτια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κοίτα λίγο τις ε, λειτουργίες μέσα στην αγορά, επίπεδο 2 και 3. Κοιτάξτε, εμείς τα κοιτούμε όλα και με το Fixing.com και τις λειτουργίες και τις επιχειρήσεις της τράπεζας είδαμε ότι υπήρχε σημαντική μείωση του κινδύνου για τις τράπεζες από το ενεργητικό επίπεδο 2 και 3 για όσους δεν γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η διάκριση. Έχουμε εδώ να κάνουμε με λογιστικά ε, πρότυπα ή έννοιες λογιστικές, ε, επιχειρήσεις δηλαδή στην αγορά στο επίπεδο 2 και 3 αυτό, αυτό σημαίνει. Σε μία λοιπόν συνολική αξιολόγηση Έχουμε 47,5 δις και με πολύ διεξοδική και εις βάθος ανάλυση των ε, ενεργητικών επίπεδου 3, κυρίως του 3, έχουμε αυτά 42,9 πιστώσεις και 49,6 δραστηριότητα στις αγορές ή συναλλαγές στις αγορές. Άρα τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, προς το παρόν τουλάχιστον. Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι το ενεργητικό επίπεδο 2 και 3 δεν είναι τοξικό ενεργητικό. Δεν είναι μη εξυπηρετούμενο. Ιδάλλως θα, το, ε, θα του επέφερε ένα πλήγμα αμέσως η αξιολόγηση από πλευράς της αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση μπορούμε εμείς να ελέγχουμε. Άρα τα κοιτάμε όλα, τα εξετάζουμε όλα, δεν ε, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία, δεν δίνουμε λιγότερη σημασία σε έναν κίνδυνο από ό,τι σε έναν άλλον, γιατί έχουμε τα μάτια μας τραβένα αλλού. Έχουμε ευρυγονική όραση. Ναι, αλλά δεν είναι ρευστά. Και είναι και μεγάλα ποσά. Ναι, βεβαίως, ε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο κύριος Τσάνη. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Άνουη, συγχωρήστε με, αλλά θα μπορέσω να συμφωνήσω με την εφορική σας διάθεση και την αισιοδοξία των ευρωπαϊκών αρχών σε σχέση με την εφαρμογή για πρώτη φορά της οδηγίας BRTD. Έχουμε ακόμα πολλά δεφιλονικούμενα και ασαφείς θέματα και βγαίνουν σιγά σιγά και οι ειδήσει. Ίσως κάποιες, επιχειρήσεις, κάποιες ε, κάποια ΜΜΕ ενημερώνονται μάλιστα καλύτερα και πιο γρήγορα από εμά, πράγμα το οποίο μας λυπεί ιδιαίτερω. Η ε, απουσία ευρωστίας της ε, Τραπεζικής Ένωση ήδη έχει καταδειχθεί. Και αναγκαστήκατε κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσετε τα γεγονότα για την ε, ρευστότητα που πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Θα ήθελα να αντιληφθώ πώς μια αρχή όπως η δική σας, που έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί στενά το ζήτημα της ρευστότητας του συστήματος του τραπεζικού των τραπεζών, θα μπορούσε να επιτρέψει τραπεζικό ίδρυμα να βρεθεί σε σχεδόν απουσία ρευστότητας μέσα στη μέση μιας εβδομάδας, κατά ημέρα εργάσιμη, με αγορές ανοιχτές και προφανώς αυτό σημαίνει ότι κάτι καλά. Και στον τρόπο της παρακολούθησης από πλευρά σας των ε, εγγυήσεων για τη ρευστότητα από την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί και η Banco Popular ε, διατύπωσε αίτημα για 40 δις εγγύησεις προς την ΕΚΤ, το οποίο αίτημα απάντησε με 3,5-4 δις ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή έδωσε 10%, το 10% από αυτό που είχε ζητηθεί. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται ξύναν τον πάτο του τσουκαλιού. Και εσείς λέτε ότι δεν καταλάβατε τίποτα. Θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Και μια γενική παρατήρηση για να ολοκληρώσω για την Τραπεζική Ένωση και το BRRD. Ε, αντί να προληφθεί το bank run, η μαζική δηλαδή άντληση ρευστότητας από τους ε, καταθέτες, φαίνεται τελικά να ε, επιτρέπεται μόνο στους μεγάλους καταθέτες ε, και επενδυτές να ξεφεύγουν με τη δυνατότητα μέσω του BRRD να ξεπούλουν τις ε, τράπεζες που βρίσκονται σε οικονομική... Παρακαλώ Που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία και που στη συνέχεια από ό,τι φαίνεται ξεπολούνται σε συνθήκες πολύ πιο ευχερείς. Όπως το Banco Santander που στην αρχή είχε προσφερθεί προς πώληση με πολύ ψηλότερο, μάλλον είχε ζητηθεί προς αγορά με πολύ ψηλότερο, μα πρόεδρε εσείς μιλήσετε 10 λεπτά, αφήστε με και να τελειώσω, με πολύ ψηλότερο τίμημα στην πρώτη πλειοδοσία και μετά ξεπουλήθηκε για ένα ευρώ. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να, γίνεται, να, να φτάνουμε σε μια συστημική κρίση χωρίς να την ελέγχουμε. Ναι, πότε γνωρίζουμε ή αν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι μπορεί να έχει μηδενική ρευστότητα ή σχεδόν μηδενική μια τράπεζα. Κοιτάξτε, τράπεζα μπορεί να χαρακτηριστεί ασθενική και τότε έχει κάθε ημερινή παρακολούθηση της ρευστότητά της ή πιθανώς ασθενική αν χαρακτηριστεί ακόμη. Και έτσι αν φανεί ότι βρίσκεται σε επικίνδυνο επίπεδο η παρακολούθηση της ρευστότητας πάει ώρα με την ώρα. Και πάλι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο ε, θέση σε λειτουργία του μηχανισμού. Μου ρωτήθηκε ήδη το ερώτημα. Απλώ όταν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ε, να δώσει η τράπεζα ρευστότητα μόνο στον πρώτο που θα εμφανιστεί, first come, first pay δηλαδή, ή όταν υπάρχει πρόβλημα ή ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα ρευστότητα, τότε δεν ενεργοποιείται ο κανονισμός, ο μηχανισμός για την αντιμετώπιση. Το BRD λέτε μπορεί να διευκολύνει το bank run. Εγώ δεν είμαι νομοθέτης. Δεν έχω σχετική αρμοδιότητα. Αλλά μπορώ να απαντήσω πως δεν το βλέπω. Το BRD στη συγκεκριμένη περίπτωση δοκιμάστηκε. Ναι, μπορούν να βελτιωθούν αρκετά πράγματα, ε, ε, μέτρα πρόορης ε, παρέμβαση σε ένα μορατόριο ασφαλώς, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία η οδηγία BRT. Ίσως όχι σε κάθε περίπτωση, αλλά στη συγκεκριμένη ναι. Για το ELA, το πρόγραμμα ρευστότητας, εγώ δεσμεύομαι από την αρχή της διάκρισης, του διαχωρισμού. Σχέση με το ELA δεν έχω. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, όσο υπάρχουν όσο υπάρχει δυνατότητα για παροχή εγγύσεως, μια τράπεζα μπορεί να ωφεληθεί από το σύστημα ELA. Ε, Και εξ όσων γνωρίζω από τα προηγούμενα χρόνια της ε, εποπτείας όταν κανείς κινδυνεύει να μην ε, μπορεί να αποπληρώσει και να χρησιμοποιήσει το χρήμα του φορολογούμενου, τότε υποχρεούται σε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο των Οικονομικών και αυτό συμβαίνει. Τον... Ευχαριστώ. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά το ρόλο της ΕΚΤ στην Σλοβενία, την πατρίδα μου. Θα τα πω γρήγορα. Όπως ε, και σε άλλες χώρες, η Σλοβενία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο της και με την συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανακεφαλαιοποίηση της Νόβα Λιουμπλιάνσκα Bank που είναι η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα πραγματοποιήθηκε και υπήρξε δέσμευση από την κυβέρνηση ότι η τράπεζα αυτή θα ε, πουληθεί έως ε, το τέλος τη φετινής χρονιάς. Πριν από λίγες εβδομάδες όμως η κυβέρνηση αποφάσισε να υπαναχωρήσει και έτσι η τράπεζα δεν θα ε, πουληθεί. Υπάρχει όμως και άλλη ιστορία από πίσω. Και αυτή αφορά την ε, διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής του Σλοβένικου Κοινοβουλίου προκειμένου να διαπιστωθεί τι τελικά ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την τόσο δυσάρεστη και δύσκολη θέση την ε, τράπεζα. Ε, έκπληκτα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ε, διαπίστωσαν ε, τα εξής. Ότι στο παρελθόν η NLB δεν χορηγούσε μόνο αμφιλεγόμενα δάνεια τα οποία οδήγησαν στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης της αλλά ότι η ίδια η τράπεζα συμμετείχε σε διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Υπήρξαν μεταφορές ενός δισεκατομμυρίου ε, ευρώ από την Ιρανική ε, ε, από Ιρανική τράπεζα, ε, γεγονός το οποίο μάλιστα αποκαλύφθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ερώτημα μου λοιπόν προς εσάς είναι το εξή. Αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως ε, βασικό καθήκον να εξασφαλίζει την ευρωστία των ευρωπαϊκών τραπεζών και καθώς η NLB είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα, γνώριζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτές τις παρατυπίες είχατε ενημερωθεί για αυτήν την περίπτωση ξεπλήματος ε, χρήματος και ποια είναι, ε, ποιος είναι ο ρόλος των εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Και τώρα που τα γνωρίζετε όλα αυτά, τι θα κάνετε. Ποιος θα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας παρακολούθησα πολύ προσεκτικά, διότι πολλά από αυτά που είπατε ε, συνέβησαν πριν αναλάβω εγώ τα καθήκοντά μου στον SSM και πριν καν δημιουργηθεί ο SSM. Όσον αφορά τη, τα μέτρα κατά της ε, νομοποίησης παράνομων εσόδων, ε, δεν είναι δική μας ευθύνη. είναι ευθύνη των εθνικών αρχών αυτό το θέμα. Πολλές φορές είναι οι κεντρικές τράπεζες ε, ή κάποια άλλη υπηρεσία εποπτείας των τραπεζών ή μπορεί να είναι και στην ίδια υπηρεσία, αλλά εμείς δεν έχουμε την ευθύνη ε, Παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Προφανώς βέβαια όταν ενημερωνόμαστε, κάτι που δεν συμβαίνει πάντοτε, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημάδι ε, κακής διαχείρισης ε, κινδύνου, κακής διακυβέρνησης, ε, κακής διοίκησης εσωτερικής. Οπότε αρχίζουμε και εξετάζουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα στοιχεία, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και βεβαίως το καταγράφουμε ως κάτι αρνητικό. Ε, στην αξιολόγηση που κάνουμε για την ε, εκάστοτε τράπεζα. Αυτά όμως μπορώ να σας πω, διότι όπως ε, σας είπα και νωρίτερα, δεν είναι δική μας ευθύνη η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το Banco Popular, γιατί τελικά αν κάνουμε μία σύνοψη όλα πήγαν καλά γιατί βρέθηκε αγοραστής αν δεν είχε βρεθεί αγοραστής, τι θα είχε γίνει. Και δεδομένης της κατανομής των στοιχείων ενεργητικού μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, αν το δει κανεί, θα καταλάβει πως στην πρώτη γραμμή διαπραγμάτευσης είχαμε τις Ισπανικές αρχές. Το ζήτημα είναι ποια θα ήταν η ενδεχόμενη ε, συνέπεια μιας ε, ε, χρεοκοπίας και για τους Πορτογάλους στην περίπτωση αυτή. Κατανοώ αυτό που μας εξηγήσατε και το γεγονός που θεωρείτε πως τέλος καλό όλα καλά, όμως εάν δεν είχε βρεθεί αυτός ο αγοραστής, τι θα είχε γίνει. Και γι' αυτό πρέπει να επιμείνω και πάλι σε ένα σύστημα ευρωπαϊκών εγγυήσεων των ε, καταθέσεων, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό δεν υπάρχει ούτε καν μία λύση τύπου ίντις και των δυνατοτήτων που έχουμε στην ΕΚΤ για να προσφέρουμε εγγύησει. Μας είπατε πως δεν είστε υπεύθυνοι για τη μάχη κατά της ε, φοροδιαφυγής. Όμως, εγώ σας έστειλα και μια γραπτή ερώτηση, στην οποία ακόμα δεν έχετε απαντήσει, για μια πρόσφατη μελέτη από την Oxfam, και που εντοπίζει τη δράση ευρωπαϊκών τραπεζών σε φορολογικούς παραδείσους. Νομικά καταλαβαίνω πως αυτό δεν αποτελεί α, τμήμα της δικής σας εντολής και της αρμοδεότητας, αλλά το γεγονός πως κάνετε υποπτία θα πρέπει να σε επιτρέπει να επαληθεύετε πώς συμπεριφέρονται οι τράπεζες και αν ανταποκρίνονται στους στόχους σταθερότητας γιατί είστε ο μόνος υπόπτη ε, για τι ευρωπαϊκέ τράπεζε. Οπότε, αν δεν το κάνετε εσείς, ποιο θα το κάνει. Και αν πείτε πως δεν είναι η δική μου δουλειά, το κάνει η Oxfam, εγώ δεν μπορώ ε, κτλ. Τότε θα πρέπει επιγόντως να αλλάξουμε την νομοθεσία και να δούμε πώς μπορούμε ε, να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Θα απαντήσω στα αγγλικά, έτσι ώστε να με καταλάβουν όλοι στην αίθουσα. Να σας πω πως καταρχήν δεν είναι πρόβλημα γιατί βρέθηκε αυτός ο αγοραστής. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίστηκε ένας αγοραστής ο οποίος αγόρασε όλη την τράπεζα και ανέλαβε όλες τις ευθύνες και όλες τις υποχρεώσεις, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και οποιοδήποτε νομικό κίνδυνο που ενδεχομένως θα ε, εμφανιστεί ε, λόγω του θέματος της ε, κεφαλαιοποίησης. Κάτι το οποίο είχε προκύψει με την ανακεφαλαιοποίηση του 2016 βάσει στοιχείων τα οποία κατόπιν προσαρμόστηκαν. Οπότε ναι, πεδίο λαμπρό για αγωγές. Παρ' όλα αυτά εμφανίστηκε ένας αγοραστής και είπε όλα δικά μου και θα αντιμετωπίσω με όλη την κατάσταση που θα προκύψει. Αν λοιπόν υπήρχε άλλη δυνατότητα, τι θα είχε συμβεί. Δηλαδή, ο αγοραστής να εμφανιστεί και να πει δεν τα θέλω όλα. Οπότε στην περίπτωση αυτή να χρειαστούμε εμείς να καλύψουμε ε, με κονδύλια τον κίνδυνο προσφυγών κατά του αγοραστή, για παράδειγμα. Ή να γίνει μια απόσπαση των πιο αδύναμων ε, τμήματων της τράπεζας, για παράδειγμα, της ακίνητης της περιουσίας και να απολυθεί το υπόλοιπο. Οπότε δεν μπορεί να τα πει κανείς ε, άσπρο-μαύρο. Πρέπει να σας πω πως το να έχει κανείς έναν αγοραστή βοηθά στο εξή, ότι ανοίγει η τράπεζα χωρίς καμία διαταραχή από τη στιγμή που αποκτήθηκε μέχρι τη στιγμή που ανοίγει τις πόρτες της. Που είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν υπήρχε καλύτερη δυνατότητα. Δηλαδή ξανά άνοιξε μέσω της εβδομάδας την επόμενη μέρα χωρίς επαναλαμβάνω ιδιαίτερες αναταραχές. Πάντως έχετε πολύ το δίκιο. Το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων λείπει. Και εδώ θα είχαμε ενδεχομένως συνέπειες, όχι απαραίτητα λόγω της ε, εμφάνισης αγοραστή για ολόκληρη την τράπεζα ή όχι, αλλά ναι, για την περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου ε, έχουν ήδη καταστήσει το σύστημα αυτό και έχουν χρησιμοποιήσει τις εγγυήσεις καταθέσεων για άλλες τράπεζες και για άλλα παρόμοια θέματα και καλύφθηκαν εκεί οι σχετικές δαπάνες. Και επειδή ήταν θηγατρικές, εάν ε, έπρεπε να μπει σε καθάριση η τράπεζα, τότε ναι, αυτό θα ήταν και πάλι αρμοδιότητα των πορτογαλικών αρχών. Τουλάχιστον μέσω του σχήματος εγγύησης καταθέσεων θα έπρεπε να αναλάμβουν δηλαδή το κομμάτι αυτό. Αλλά σίγουρα δεν θα ήταν κάτι τέτοιο μια ιδανική λύση και ελπίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων θα ισχύσει θα εφαρμοστεί. Έχουμε όμως αυτή τη στιγμή και τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό και το SRB και όλες τις δυνατότητες να συνεργαστούμε με τις πορτογαλικές και τις ισπανικές αρχές που έδειξαν φοβερό πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να έχουμε τέτοιου είδους πετυχημένα αποτελέσματα. Εγώ σήμερα έμαθα πως μου στείλατε τον Απρίλιο μια ερώτηση. Εμείς λάβαμε την ερώτησή στις 8 Ιουνίου και γι' αυτό δεν έχετε πάρει εσείς ακόμα απάντηση. Από τις 8 Ιουνίου μέχρι σήμερα οι συνεργάτες ε, μου δούλεψαν την απάντηση και έχω ένα σχέδιο ε, το οποίο θα σας στείλω και θα το κοιτάξω γύρω από τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να φτάσει. Να σας πω πως ως πολίτης Μοιράζομαι απόλυτα την άποψή σας, συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή σας πως όλα αυτά ε, για την καταπολέμηση της ε, ε, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, της ξεπλήματος θα έπρεπε να διώκονται και δεν αντιμετωπίζομαι καμία συμπάθεια ανθρώπους ή οργανώσεις που χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους έτσι ώστε να μην συνεισφέρουν αυτό το οποίο τους αντιστοιχεί στην κοινωνία τους, στη χώρα τους, στην περιφέρειά τους. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε τέτοιου είδους αρμοδιότητα και δεν είναι επειδή δεν έχουμε αρκετούς πόρους, αλλά θα σας έλεγα το εξή. Είναι θέμα νομοθέτη ή κοινοβουλίου αν θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, καταπολέμησης νομοποίησης παράνομων εσόδων και νομίζω ότι θα μας βοηθούσε γιατί έχουμε αρκετές μικρές χώρες που αυτή τη στιγμή πληρώνουν υψηλό τίμημα ε, για το σύστημα της αντίστοιχης τραπεζικής συναλλαγής. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 εταίρους και 8 τράπεζες, 25 συνολικά είμαστε, που προσπαθούν να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος. Δεν βρίσκεται στο κομμάτι αυτό της εποπτείας βέβαια, αλλά νομίζω πως για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου αρμοδιότητε θα έπρεπε να έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο που θα είναι σαν ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Οπότε για ένα νέο σύστημα κατά τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων νομίζω ότι θα έπρεπε κάτι να γίνει. Ο Γκαμπριέλ Μάτο. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω με τον Banco Popular γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ε, με ανησυχεί. Μικροκαταθέτες, μικροεπενδυτές που λένε κάπου κάναμε λάθο. Και ανησυχώ. Και ανησυχώ γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θίγεται η ίδια η αξιοπιστία του ενιαίου ποπτικού μηχανισμού. Και πρέπει να σας πω ότι και η δική σας απάντηση με άφησε ε, ανησυχώ, γιατί βλέπω να έχουμε κάποιο είδους αυτοπεποίθησης ε, και αυτοικανοποίησης από το γεγονός που συντάξει ξανά άνοιξε τις πόρτες χωρίς να μπουν δημόσια κονδύλια. Άρα είχαμε μια μεγάλη επιτυχία και αυτό αποδεικνύει πως η ισπανική οικονομία είναι ισχυρή. Εντάξει, το δέχομαι αυτό. Ε, η τράπεζα τα αντιμετώπισε. Αλλά δεν μπορεί, κάπου κάναμε λάθο. Συ, ε, ε, αν έχουμε λοιπόν ε, πέρσι μια τράπεζα που περνά κάθε δοκιμή και κάθε δοκιμή λέει μπορεί να πετύχει ε, καλά αποτέλεσματα ακόμα και στα αντίθετα σενάρια και ξαφνικά βρισκόμαστε εκεί που είμαστε, τι έγινε με τα stress test. Γιατί δεν το βρήκαν, γιατί δεν το αποκάλυψαν και είπαν ότι ναι, εντάξει, είχαν και τα κακά σενάρια και τα λοιπά, αλλά συγγνώμη, αν συνέβαιναν όλα αυτά, ε, γιατί τελικά καταλήξαμε εκεί που βρεθήκαμε. Και τέλος θα ήθελα να μου πείτε, εάν κάπου κάναμε λάθος, ποιο είναι το δίδαγμα το οποίο αποκομίζουμε. Γιατί εδώ έχουμε τον πρώτη εφαρμογή του συστήματος και το σύστημα είναι καλό, το πιστεύω, αλλά κάπου κάναμε λάθος κάπου κάναμε λάθο ή όχι. Πιστεύετε εσεί ότι τα πήγαμε θαυμάσια. Σε εποπτικό επίπεδο. Δεν μιλώ για κάτι άλλο. Σε εποπτικό επίπεδο. Δεν κάναμε κανένα λάθο. Και θα ήθελα να μου πείτε εάν οι επόπτε, για παράδειγμα, δεν έχουν τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου καταστάσει. Ή λείπουν τα εργαλεία ή έχετε τα εργαλεία και δεν τα εφαρμόσατε σωστά. Ποια είναι η απάντηση. Και τέλο θα θέλω να μου πείτε εσείς θεωρείτε πως λειτουργήσαν σωστά οι μηχανισμοί δράσης για τις ταπεζικές κρίσεις, για προβλήματα ρευστότητας. Το έχουμε συζητήσει πολύ. Έχουμε μηχανισμούς. Λειτουργήσαν ή όχι. Γιατί εμείς δεν μπορώ να σας πω ότι αισθανόμαστε ήσυχοι πως κάτι αντίστοιχο δεν θα ξανασυμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι μου λέτε ότι το κλείσιμο μιας τράπεζας είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. έχουμε κηρύξει ως ε, ε, τράπεζα που κινδυνεύει να ε, χρεοκοπήσει μόνο μία. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο προστατεύσαμε τα χρήματα των καταθετών τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν λέω ότι είναι μια εύκολη, μια λαμπρή ή μη επώδυνη απόφαση αυτή, αλλά δυστυχώς να σας πω Ελπίζω και την επόμενη φορά το ίδιο να κάνουμε. Να μπορέσουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι την επόμενη μέρα η τράπεζα θα ξανανοίξει χωρίς να χάσει κανείς τα χρήματά του. Και το μήνυμα που είχα λάβει μέχρι στιγμής δεν ήταν ποτέ ότι δεν πρέπει ποτέ να κηρύξουμε ως πτωχευμένη μια τράπεζα ή ότι δεν πρέπει ποτέ μια τράπεζα να κλείνει. Δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ αυτό. Σκεφτείτε την βλάβη μάλιστα που θα προκαλούσε κάτι τέτοιο σε όλες τις άλλες μεγάλες ισχυρές τράπεζες ε, όταν υπάρχει μια υπερπροσφορά, υπερπροσφορά τραπεζικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα ήταν σαν να διατηρούμε τεχνητά όλες τις τρα... στη ζωή όλες τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτό θα ήταν πρόβλημα. Όχι το να έρθουμε μία φορά στα τρία χρόνια και να κηρύξουμε επιτοχευμένη μία τράπεζα και έχοντα εξασφαλίσει μάλιστα ότι κανεί δεν έχασε τα χρήματά του και ότι η τράπεζα άνοιξε την επόμενη μέρα. Διδάγματα. Δύο νομίζω ότι είναι τα διδάγματα. Πρώτον, οι επόπτες πρέπει να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες προκειμένου να εξασφαλίζουν έγκαιρη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Νομίζω ότι κάθε δάνειο που δεν εξυπηρετείται θα πρέπει να αντισταθμίζεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ υψηλά, υψηλές αναλογίες CET ε, και αυτές βασίζονται σε χαμηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μόλις όμως αρχίσουν να αντιμετωπίζουν, αντιμετωπίσουν την κατάσταση έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα, θα αντιμετωπίσουμε καινούρια προβλήματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε την, ε, ε, ε, την ρευστότητα και την, τον υγιή, την ευρωστία όλων των τραπεζών. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε στο, στο μέλλον. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα καλύπτονται από, από μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται έγκαιρα για την αντιμετώπιση αυτών των δανείων και όχι από ε, μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν στο να μην υπάρχουν καθόλου απώλειες. νομίζω ότι δεν είπατε ποτέ ότι το πρόβλημα είναι το κλείσιμο μιας τράπεζας. Να σας πω ότι χαίρομαι που δεν έκλεισε η τράπεζα, όχι γιατί ήταν επιτυχημένη η εποπτεία, όχι, αλλά γιατί έδειξε πως είναι στεναρή η ισπανική οικονομία. I don't think you, you need to reply unless you wish. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσετε, εκτό αν θέλετε. Όχι. Ε, εν πάση περιπτώσει, κανεί δεν είπε εδώ ότι το πρόβλημα είναι η εξυγίανση μια τράπεζα. Το πρόβλημα είναι ότι έγινε με αυτόν τον τρόπο τόσο απότομα ε, και ότι ε, ακούγαμε για υπερβολικά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την τράπεζα. Ευχαριστώ, είμαι εδώ. Θα συνεχίσουμε με τον Banco Popular. Μας είπατε πως λύθηκε χωρίς να δημιουργήσει τριβές. Νομίζω πως δεν γνωρίζετε πως ο επόπτης αγορών αυτή τη στιγμή ε, απαγορεύσε το short selling ε, στην Ισπανία και η αγορά έζησε πολύ δύσκολες ημέρες μετά από αυτή την απόφαση. Οπότε όντως κάποιες τριβές δημιουργήθηκαν. Και να σας πω πως ε, το, η Banco Popular δεν είχε μόνο πρόβλημα ρευστότητα, γιατί αν ήταν μόνο αυτό, έχουμε τα εργαλεία και είναι επαρκή για να το αντιμετωπίσουμε. Το ζήτημα είναι ε, πώς μας παραξενεύει πώς δεν χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία αυτά. Γιατί είπατε πως μπορείτε εσείς να επέμβετε εγκαίρως και θεωρήσατε πως δεν χρειάστηκε λόγω του κόστου που είχε αξιολογηθεί και πως τελικά ουσιαστικά οδηγηθήκαμε σε μια λύση σαν αυτή στην οποία καταλήξαμε. Άρα λοιπόν, πώ είναι δυνατόν μια τράπεζα όπω η Banco Popular να μείνει χωρί ενέχειρα και εγγύηση έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα. Πώ είναι δυνατόν η διαδικασία με τα μέτρα για να προσφέρει ρευστότητα σε μη ρευστέ τράπεζε δεν χρησιμοποιήθηκε επαρκώ. Νομίζω πω προφανέστατα υπήρχε πρόβλημα φερεγγιότητα και το ζήτημα είναι, μέσα σε αυτό το πακέτο δράσεων πρέπει να δούμε αν ο ε, μηχανισμός, ο ενιαίος υποπτικός μηχανισμός κατάλαβε πού το έχασε και αν μπορείτε εσείς να κάνετε ένα απολογισμό και να πείτε τι συμβαίνει, γιατί ε, όταν ε, κάναμε τα τεστ ε, η Banco τα πέρασε. Τώρα, για την έκθεση σύμφωνα με την οποία εκινήθηκε η διαδικασία θέλουν να δημοσιευθεί, να δούμε πώς ποσοτικοποιήθηκαν αυτές ε, ε ανάγκες σε 2 με 8 δις που αποφασίστηκαν. Θα ήθελα παρακαλώ αυτά να τα διαβάσουμε. Και επίσης μας είπατε πως εσείς δεν έχετε σε όλα τα θέματα φωνή. Όμως για μας υπάρχει πρόβλημα εποπτείας γιατί για κάποιο λόγο οι ισολογισμοί δεν εμφανιζόντουσαν σωστά και αυτό δεν το είπε κανείς. Είχε μπει και προηγουμένως σε διαδικασία πώληση και πρέπει να σας πω ότι αυτού του είδους οι αγοροπολισίες δημιουργούν αυτόν τον ηθικό κίνδυνο, αυτό το moral hazard για την περίπτωση που κάποιοι θεωρήσουν πλέον ότι είναι καλύτερο να περιμένουν να αγοράσουν αφού μπει σε διαδικασία λύσης παρά να αγοράσουν προηγουμένως έτσι ώστε να αποφύγουν κάποιες ενδεχόμενες αγωγές για απόλυση ζημίες. Οπότε αυτό είναι ένα κακό προηγούμενο. Ε, μου θέσατε πολλές ερωτήσεις που για να τις απαντήσω θα έπρεπε να παραβώ τους όρους εμπιστευτικότητας. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα για την κατάσταση της ε, τράπεζας. Όσον αφορά το ζήτημα ρευστότητα, μπορώ να σας πω ότι εκτός όσων γνωρίζω, γιατί δεν είναι ε, στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου, ε, σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει ο ELA αλλά είναι εθνική αρμοδιότητα. Το κράτος πρέπει να ζητήσει ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για εθνικό κίνδυνο και ότι, ε, και ότι μάλιστα βρίσκεται στα αρχικά του στάδια. Ανάλογα και με τα ποσά που εμπλέκονται κάθε φορά. Όσον αφορά τα σφάλματα κατά την εποπτεία. Ε, φυσικά και θα κάνουμε νεκροψία. Είναι προφανές. Ε, και μάλιστα θα είναι και πολύ προσεκτική η διαδικασία αυτή. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν, υπάρχει μια συνύπαρξη στοιχείων που παραγόντων που οδήγησαν την τράπεζα στην χρεοκοπία. Θα δούμε και από την ανάλυση μας αν κάναμε ό,τι μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε και θα δούμε θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Για, το, για αυτό τον ηθικό κίνδυνο για τον αγοραστή πρέπει κανείς να το δει και από τις δύο σκοπιές του αγοραστή και του πολιτή. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν θέλω να συζητήσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αντίσταση να αγοράσει κανείς υπό τις ε, συνήθεις, τις κανονικές συνθήκες προέρχεται από τον ε, πολιτή γιατί βλέπει ότι δεν, δεν παίρνει την τιμή που θα ζητούσε. Γιατί η Banco Popular είχε ανακοινώσει στην αγορά ότι θέλει να, να πολιθεί ε, και αυτή η πληροφορία ε, μάλιστα βοήθησε και στο να υποβληθούν και συγκεκριμένε προτάσεις από άλλες τράπεζες ε, και έτσι επιταχύνθηκε η διαδικασία. Ωστόσο, ο πολιτής δεν αποφάσισε να πουλήσει τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο τελικά στην τιμή που του προσέφεραν οι πιθανοί αγοραστές. Είναι λίγο σαν το θέμα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, ξέρω ότι πολλές φορές ε, η πώληση δεν γίνεται γιατί η τιμή δεν είναι στο σωστό επίπεδο. Αν εγώ πουλήσω το διαμέρισμά μου, το διαμέρισμά μου τις περισσότερες φορές αυτό που πιστεύω είναι ότι η αξία είναι υψηλότερη γιατί μου αρέσει, γιατί έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη ζωή μου σε αυτό κτλ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις τράπεζες. Ε, πας να πουλήσεις μια τράπεζα, έχεις μια εικόνα για το που θα, ε, για το που θα ε, έπρεπε να ε, κάτσει μπάλα αλλά αν δεν βρεις αγοραστή που να σου δώσει αυτά τα λεφτά τότε κάθεσαι εσύ και το περισσοκό σου στοιχείο. Οπότε καλό είναι να γίνεται αυτή η διαδικασία αρκετά έγκαιρα προκειμένου να μην αντιμετωπίζεται αυτός ο ηθικός κίνδυνος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με εντυπωσιάζει πραγματικά αυτή η αυτοπεποίθησή σας ότι πάντοτε τα πράγματα στις αγορές ήταν ε, ιδανικά. <laughs> Κύριε Φίπνερ, Κοιτάξτε, ε, δεν ξέρω πότε θα σας ξαναδώ, κυρία Πρόεδρε, γι' αυτό θέλω να διατυπώσω ερώτηση για την αναθεώρηση της ΕΣΑ. Ε, αναφέρατε νωρίτερα με μια ε, έκφραση, ανακούφιση θα έλεγα, ότι δεν ψηφίζετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, ναι, αλλά ίσως κάποιοι να θεωρούσαν ότι θα ήταν σκόπιμο να έχετε και δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι συμμετέχετε ουσιαστικά στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Επίσης είναι πολύ η θεωρητική της οικονομίας που θα λένε ότι θα πρέπει η ΕΤΑ να έρθει πιο κοντά στην ΕΚΤ, ενώ κάποια άλλη μια άλλη σχολή, ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο. Κάποιοι άλλοι μιλούν για έναν σταθερό διαχωρισμό μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΑ. Εσείς έχετε κάποια θέση σε αυτό προς τα πού θα θέλατε να πάνε οι υπηρεσίες προς το μέλλον. Ο Μοργκάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις τελευταίες ανταλλαγέ απόψεων ε, με την Επιτροπή μας, κυρία Νουή, Έγιναν ε, αναφορές σε θέματα που έχουν να κάνουν ε, με την Τραπεζική Ένωση, βεβαίως πολλές φορές με ιδιαίτερη έμφαση σε ρυθμιστικές ε, διατάξεις. Αυτή την εβδομάδα, παραδείγματι, θα κάνουμε συζήτηση για τροποποίηση του CRR, για τις CRR της οδηγίας, για ένα μεταβατικό καθεστώς για το IMIFRS e σε μια νέα προσέγγιση, όχι στατική. Ε, το αναφέρω αυτό γιατί ίσως ε, θα ήταν σκόπιμο να κοιτάξουμε να περιορίσουμε την εισαγωγή της λογιστικής λογικής σε σχέση και με τις ΗΠΑ που θα τεθεί σε ε, ισχύ το 2020. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια προληπτική αντιμετώπιση του χρέους, του κρατικού χρέους που διακρατούν τράπεζες με παρακολούθηση της, του τρόπου άσκησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκριτικό μειονέκτημα για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Δεδομένου ότι η αγορά θα αντιδράσει σε αυτό το άνοιγμα. Και επίσης έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας με ανάπτυξη ασθενική και χωρίς τη δυνατότητα τους τίτλους ε, που έχουν προβλήματα να τους ε, αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε. Με μη εξυπηρετούμενες πιστώσεις τόσο για τις Ισπανικές και τις Ιταλικές τράπεζες που οδήγησαν στην πρώτη εκαθάριση της Banco Popular αποδεικνύεται ότι το BRRD δεν είναι άμυρο προβλημάτων. Γι' αυτό λοιπόν τη με και σας ρωτώ, μήπως θα έπρεπε πρώτα να αναπτύξουμε περισσότερη εμπειρία σε σχέση με τους υφιστάμενους κανόνες. Και αν συμφωνείτε ότι οι προτάσεις για τροποποίηση θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες ε, σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα και την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου πρώτα να απαντήσω στην παρατήρηση του Προέδρου για την υπερβολική μου εμπιστοσύνη προς τις αγορές. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Για ορισμένα πράγματα ιδιαίτερος δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις αγορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υψηλές τιμές στην κεφαλαιοποίηση των αγορών, που ήταν το πρόβλημα άλλωστε που εντοπίστηκε και σε ένα βαθμό εξηγεί και το γιατί η τράπεζα δεν θέλησε να απολυθεί σε μια πιο πρόσφορη τιμή. Γιατί θεώρησε το Συμβούλιο ότι υπήρχε κίνδυνος να μην πολυθεί η τράπεζα στο ύψος που ήθελε. Γι' αυτό λοιπόν δεν εμπιστεύομαι τις αγορές. Άλλες φορές τα πάνε καλά, άλλες λιγότερο. Και όχι, δεν αισθάνομαι ανακούφιση που δεν ψηφίζω στην ΕΤΑ. Εγώ απλώς νομίζω ότι θα έπρεπε στην ΕΤΑ να είναι πιο ισχυρή η φωνή της Ευρώπης. Ο Ανδρέα Ενρίε παραδείγματι δεν ψηφίζει. Αυτό με ξεχνιάζει. Και είναι σφάλμα. Ευρωπαϊκή ε, φωνή δεν υπάρχει. Ελπίζω στο τέλος οι εθνικές φωνές και ψήφοι γύρω από το τραπέζι της ΕΚΤ να συμπληρωθούν από μια ευρωπαϊκή. Δεν ξέρω πότε, αλλά εν θα πρέπει να ισχυθεί η θέση της Ευρώπης με πρώτη την ε, ψήφο του Ανδρέα Ενρία. Τώρα, ποιες αλλαγές από το Brexit για την ΕΤΑ. Δεν ξέρω να σας πω. Αλλά έχει μάλλον ρυθμιστικό ρόλο η ΕΤΑ. Προσπαθεί να εναρμονίσει οδηγίες, ε, να καταστήσει επιχειρησιακή την νομοθεσία, πράγμα το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, γιατί να το κάνει η ίδια η ΕΜΠΑ, θα πρέπει να το πράξουμε εμείς και είναι βαρύ έργο. Εν και των εθνικών επιλογών. Και άρα ως ρυθμιστής, περισσότερο ρυθμιστικού ε, χαρακτήρα αρχή η ΕΤΑ έχει ασφαλώς καλύτερο ρόλο από μας σε αυτό. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άμεσης υλοποίησης της νομοθεσίας πάντως. Ε, εάν δεν ψηφίζονται αλλαγές ε, ταχύρυθμες, των προτάσεων θα ε, προχωρούσαμε σε άμεση εφαρμογή του ΕΦΑΡΕΣ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό το οποίο ψήφισε μην προχωρήσουμε σε άμεση υλοποίηση. Αυτό αναφέρεται στο κείμενο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ναι, ε, μια σταδιακή εισαγωγή του συστήματος, αλλά αυτό θα πρέπει να, αυτή η σταδιακή εισαγωγή θα πρέπει να αφορά μόνο την, ε, τον πρώτο κλειδανισμό από την εισαγωγή της νομοθεσίας, το CT1 δηλαδή. Αυτό πρέπει να δούμε ως phase-in. Όμως, στο διακή εισαγωγή κάθε μέτρο που έχει ανακοινωθεί εδώ και τόσο καιρό δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να ε, προετοιμάσουμε τον κόσμο με λιγότερη έκθεση. Θέλουμε με τρόπο ρεαλιστικό αλλά πάντα φιλόδοξο να διαμορφώνουμε αυτή την, ε, αυτό το περιβάλλον, αλλά δεν θέλουμε και να ε, σορευθούν βάρη ε, για τις τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ντανιέλ Νουή, λέει ο πρόεδρος. Εντατική, πολύ εντατική η ανταλλαγή. Απόψε, αλλά βέβαια και τα θέματα που είχαμε ήταν πολύ περίπλοκα. Και πρέπει να πω ότι για το θέμα αυτό των πιθανών ελλείψεων, σε αυτό διαφωνούμε, στην εποπτεία ασφαλώς θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Και εμείς ως Κοινοβούλιο να τα ξαναπούμε πιο προσεκτικά, να αντιληφθούμε καλύτερα την κατάσταση, γιατί ασφαλώς θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πώς γίνεται η δουλειά στο μέγιστο βαθμό, ότι στο μέγιστο βαθμό αξιοποιούνται τα εργαλεία που υπάρχουν. Αν δεν αρκούν τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να ε, δημιουργηθούν νέα. γιατί ε, ας το πω έτσι έχουμε ε, υπολοιπόμενο του αρίστου πλαίσιο και λειτουργία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα συνεχίσουμε την επικοινωνία και γραπτός αλλά και σε άλλες συνεδριάσεις για να αντιληφθούμε καλύτερα τι ε, λειτουργήσε σωστά και τι λειτουργήσε λιγότερο σωστά σε αυτή τη διαδικασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών της Μάλτας, τον Εντουάρ Σκυπλούνα. Καταρχήν, να σας δείσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά έγινε μια εξαιρετικά έντονη ακρόαση με την πρόεδρο του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού. Χρησιστήκαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε φανταστεί. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ που είχατε την ευγένεια να δεχτείτε την πρόσκλησή μας έτσι ώστε να κλείσουμε ε, την Προεδρία της Μάλτα, στα θέματα της δικής Επιτροπής με αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας να ξεκινήσω λέγοντας πως θέλω να σας συγχαρώ και εσάς και την Προεδρία της Μάλτας γιατί πιστεύω πως στα δικά μας θέματα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Και πρέπει να σας πω πως είχατε και την προεδρία ε, πολλών συναντήσεων ε, τριμερούς διαλόγου Πέντε φάκελοι έκλεισαν, ξέρετε, την τιτλοποίηση, τα στατιστικά προγράμματα, ε, τα επενδυτικά κεφάλαια κινδύνου, όπως επίσης και μεγάλη πρόεδρος σε άλλα θέματα, ε, το ΕΦΣΥ, το ξέπλυμα χρήματος. και για τους λόγους αυτούς θα ήθελα και πάλι να σας συγχαρώ. Ήταν εξαιρετική η προσπάθεια που κάνατε και εξαιρετική η συνεργασία μαζί σα και πρέπει να σας πω πως πετύχατε πολλά για τους φακέλους, ο οποίους συζητήσαμε και ευρύτερα σε όλες τις προσπάθειες που κάνατε, έχοντας την Προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία προχώρησαν, για παράδειγμα, στο χώρο της φορολογίας. Θα ήθελα να επενδυμίσω λοιπόν στους συναδέλφους πως η σημερινή ανταλλαγή απόψεων εστιάζει στα θέματα της Μαλτέζικης Προεδρίας και όχι ε, τα θέματα της, τα εσωτερικά της Μάλτας. Και γι' αυτό θα σας δώσω τώρα το λόγο για να μας παρουσιάσετε το έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ πάντα είναι χαρά να έρχεται κανείς στην Επιτροπή ΕΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τονίσω που σημειώσαμε πρόοδο στην δική μας Προεδρία, τουλάχιστον στα βασικά θέματα που είχαμε στη δική μας ημερήσια διάταξη και να εστιάσω σε θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σκαριά και φτάνουν στο τέλος θα μπορούσαμε αυτά ας πούμε, να τα δούμε σε ερωτήσει οι οποίε θα ακολουθήσουν. Να σα πω πω γενικότερα, όπω και ο πρόεδρο, είμαι πολύ ικανοποιημένο. με τα όσα πετύχαμε με τις προτεραιότητες, με την ε, Ένωση Αγοράς Κεφαλαίων, με τα θέματα φρολογίας. Είχαμε μερικά πολύ θετικά αποτελέσματα και θεωρώ πως προοδεύουν και κάποια άλλη φάκελοι με ταχύ ρυθμό και ελπίζω πως και πριν το τέλος του μήνα κάποιοι από αυτούς τους φακέλους ενδεχομένως θα κλείσουν ε, μέχρι τότε. Ξέρετε ποιο είναι το υπόβαθρο, είναι η οικονομική κατάσταση που μας περιβάλλει, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, εκεί βρισκόμαστε και με χαρά βλέπουμε πως ενισχύεται η ανάκαμψη. Αυτό μας είπε και το Eurogroup ε, και στο ECOFIN η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτή η ανάκαμψη έχει στέρεες βάσεις και καλύπτει πολλούς κλάδους και όχι μόνο συγκεκριμένους άρα οι οικονομίες μας ήταν ανθεκτικές και η αβεβαιότητα έχει καμφθεί ε, μια και κάποιοι από τους πολιτικούς κινδύνους που διαβλέπαμε δεν υλοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Προκλήσεις γιατί θέλουν μακροπρόθεσμη ε, και ευρύτερη πρόοδο και ανάπτυξη. Και βεβαίως αύξηση και της προσφοράς και της ζήτησης. Και εκεί εστιάσαμε στη δική μας Προεδρία. Δηλαδή, το να οδηγήσουμε το Συμβούλιο προς το χώρο της, του συντονισμού της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, της ε, νομοθεσίας για τα χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά και την Ένωση, την Τραπεζική Ένωση, και την Κεφαλική Ένωση και να σας πω τι κάναμε με τα κράτη-μέλη και για το συντονισμό της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής αυτών. Να σας πω πως το Μάρτιο εγκρίναμε τις συστάσεις του 17 για το χώρο του ευρώ. Η υιοθέτηση αυτή ακολούθησε τις επικοδομητικές και ανοιχτές συζητήσει που έκαναν οι υπουργοί μεταξύ τους και την έγκριση, έλαβαν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι συστάσεις απευθύνονται με ισορροπημένο τρόπο στα πολλά θέματα πολιτικής που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τις ανακράτους συστάσεις του 2017 που εγκρίθηκαν από το Eurogroup και το COFIN την περασμένη εβδομάδα και επισήμως θα εγκριθούν από το Συμβούλιο μέσα στον Ιούλιο. Για τη δημοσιονομική πολιτική τα κράτη-μέλη επέλεξαν να μην ποσοτικοποιήσουν εξάντε ε, την δημοσιονομική ε, πολιτική που θα ακολουθήσουν στο χώρο του ευρώ, γιατί η πρακτική εφαρμογή έτσι καλώς δεν θα ήταν απλή με το τρέχον νομικό πλαίσιο. Όμως, πετύχαμε συνένεση και είπαμε πως μία ισόρροπη στήριξη της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή ζωή σημαίνει μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ανακράτως. Και αυτό το είπαμε στο τελευταίο στην τελευταία συνάντηση του Eurogroup όπου ακούσαμε και τις προβλέψεις του Δουνουτού όπως επίσης και ε, τα όσα έχει στο άρθρο 4 της εκθεσής του. Τα κράτη-μέλη που βρίσκονται ε, σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, έχουν ε, κληθεί να ανοίξουν τις επενδύσεις και τα κράτη-μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν υψηλότερο δημόσιο χρέος θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημοσιονομική εξυγίανση ευθυγραμμιζόμενη με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες εν ώψη των σπάνιων δημοσίων πόρων είπαμε πως θα πρέπει να επιταχύνουμε την εξέβρεση ε, κάποιας δυνατότητας περικοπής ε, έτσι ώστε ε, να, να μην στηρίζουμε τόσο πολύ τις άμεσες δαπάνες, αλλά να δούμε μακροπρόθεσμα θέματα κεφαλαιοποίησης. Να σας πω πως τα δημόσια χρέη αυτή τη στιγμή σταθερά μειώνονται και αυτό ήταν εξαιρετικά θετικό γιατί για την Πορτογαλία και την Κροατία αποφασίσαμε πως δεν χρειάζεται μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει κάτι το αντίστοιχο για την Ελλάδα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά θετικό. Και οι χρηστέ δημοσιονομικέ πολιτικέ είναι ένα κομμάτι τη αφήγηση. Και στι συστάσει είπαμε πω θα πρέπει επίση να προχωρήσουν οι δαρθωτικέ μελέτε που εξυγχρονίζουν τι οικονομίε μα και που μα κάνουν πιο ανταγωνιστικούς γιατί βασίζονται σε αύξηση τη παραγωγικότητας. Και με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουν σε μια ανάπτυξη που θα του συμπεριλαμβάνει όλου. Και αυτό βεβαίω πρέπει να γίνει με διαφοροποιημένη προσέγγιση ανακράτω τα θετικά προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη και το γεγονό πω οι δημοσιονομικέ συνθήκε μοιάζουν πολύ ενθαρρυντικέ, προσφέρουν αυτή τη στιγμή μια μοναδική, ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρία με κάποιε σφαιρικέ πολιτικέ που θα μα κάνουν πιο ανθεκτικού και θα είμαστε πιο έτοιμοι για μελλοντικέ ε, και νομίζω ότι εκεί μα οδηγεί και το κοινό μα συμφέρον. Και ε, μέσω τη ταχύα συμφωνία που πετύχαμε τον Ιανουάριο στην αρχή τη Προεδρία μα για τι διευθυντικέ ε, ε, και το σχετικό πρόγραμμα, μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη θα μπορούν πια να έχουν αυτή την εξατομικευμένη στήριξη για τις ε, μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν. Η Προεδρία μας το Μάρτιο οργάνωσε και μια συζήτηση μέσω του ΕΚΟΦΗΝ με το Συμβούλιο για τα κράτη-μέλη και για το πώς τα έχουν πάει στο παρελθόν με την εφαρμογή των ε, ε, συστάσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να αυξήσουμε την πίεση στην ε, δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Φορολογία τώρα. Να σας πω πως η δίκαιη φορολόγηση είναι μια δίκαιη ανησυχία που διακατέχει τον Ευρωπαίο πολίτη και χαίρομαι που καταφέραμε να προχωρήσουμε αυτούς τους έξι μήνες. Στις 29 Μαΐου και μετά την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμείς εγκρίναμε μια τροπολογία για την οδηγία για την φοροαποφυγή. Εδώ καλύπτουμε τους κανόνες για την φοροαποφυγή μέσω μη ε, κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνουμε δηλαδή ένα παράθυρο από την προηγούμενη νομοθεσία έτσι είναι η 882 αντεντουμένα και πρέπει να σας πω πως ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το 2019 για να έχουμε μια πλήρη εφαρμογή. Πάντως έχει δοθεί χρόνος και νομίζω πως αυτά τα δύο νομοθετικά έργα, είτε μεμονωμένα είτε συνδυασμένα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είναι σημαντικά και θα μειώσουν αυτές τις προσπάθειες που γίνονται φορο, την αφοροαποφυγή και τις σχετικές πρακτικές από τις επιχειρήσεις. Πριν από μερικές εβδομάδες το Συμβούλιο επίσης κατέληξε σε γενική προσέγγιση για την ε, ε, προτινόμενη για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών λόγω διπλής φορολόγησης έτσι ώστε να υπάρχει φορολογική βεβαιότητα για όλους τους παίκτες. Το Συμβούλιο περιμένει και την γνωμοδότηση, σχετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συζητήσει για τις ε, ε, εκκρεμής προτάσεις, τα e-publications και το μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης, όπως επίσης το πακέτο για την ηλεκτρονική συναλλαγή και τον ΦΠΑ, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Συμβούλιο, τρέχουν και είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό που χρειάζεται να σας το πω εδώ, αλλά εκεί βρισκόμαστε ακόμα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά περίπλοκα, το καθένα ξεχωριστά, γιατί ε, χρειάστηκε να δοθούν κάποιες εγγυήσεις έτσι ώστε και το πακέτο για το ηλεκτρονικό εμπόριο να ε, προχωρήσει ομαλά και τελικά βρήκαμε όλες τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και το ίδιο ισχύει και για τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ, δηλαδή κάποιες εγγυήσεις πως δεν πρόκειται αυτό να διασπαρεί και δεν θα διαδοθεί πέραν ε, του πιλωτικού ε, project από το ένα κράτος στο άλλο. Δυστυχώς όμως παρόλα αυτά τη τελευταία στιγμή δεν καταφέραμε να πετύχουμε την πολιτική έγκριση έτσι ώστε αυτό το πειραματικό ε, πιλωτικό σχέδιο να εφαρμοστεί. Και απογοητεύτηκα γιατί κάποιες χώρες το χρησιμοποίησαν ως τρόπο για να μπλοκάρουν το πακέτο για τις ηλεκτρονικές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, κάτι το οποίο επιθυμούσαν πολλά κράτη-μέλη. Αλλά σφανούμε θετικοί και αισιόδοξη ότι αυτό θα ξεπεράσει τους κοπέλους και θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Αργότερα ίσως το περιβάλλον είναι πιο κατάλληλο και για τα δύο αυτά νομοθετήματα. Είμαι αισιόδοξο ότι η Εστονική Προεδρία θα καταφέρει να χρησιμοποιήσει τα όσα οικοδομήσαμε, γιατί είναι όριμα έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά και να εγκριθούν και επισήμως στο Συμβούλιο. Για το FC2, το επενδυτικό δηλαδή αυτό το ταμείο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ξέρετε πως είναι κάτι που μας αφορά ιδιαίτερα, είναι ένα είδος επενδύσεων μεγάλου μεγέθους, μεγάλης διάστασης που είναι απαραίτητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, λειτουργεί. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε πια για σχέδιο, αλλά για κάτι το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε και γι' αυτό τρέχουν συζητήσεις ε, για την επόμενη φάση. Χαίρομαι που καταφέραμε να φτάσουμε στη φάση του τριμερούς διαλόγου για το θέμα αυτό και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκτείνει ε, το ΕΦΣΥ μετά από τη σύμφωνη ε, ε, άποψη στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το μηδέν και το προωθήσαμε. Βεβαίως τώρα χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τρεις καλή συζητήσεων και έχει ε, νομίζω μπει στο πρόγραμμα και ακόμα ένας γύρος αυτή την εβδομάδα. Έχοντας κοιτάξει τον ε, φάκελο, πιστεύω πως θα βρούμε συμβιβασμό για κάποια από τα ζητήματα τα οποία έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία δικαιολογούνται. Βεβαίως, εδώ εκφράζω τη θέση του Συμβουλίου της χώρας μου. 27 κράτη-μέλη υπάρχουν και νομίζω πως θα πρέπει να απηχήσουμε τη θέση όλων και γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται περισσότερος χρόνος, γιατί δεν είναι για όλους τόσο απλό και λογικό όσο φαίνεται σε κάποιους. Για το ΕΦΣΙ πάντως να σας πω πως για τη χρηματοδότηση υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, όπως επίσης και για θέματα που άπτονται του προπολογισμού. Εδώ έχουμε τις συνέπειες του Brexit κτλ. Οπότε δεν είναι εύκολα. Αν μείνω στο θέμα των επενδύσεων, να σας πω πως πιστεύω πως το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ακόμα στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ε, ΕΤΕ και του, της εντολής εξωτερικού δανεισμού που έχει η μετανάστευση μια πρόκληση. Δεν θα εξαφανιστεί. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεων μας. Γιατί έχουν σημασία. Και για μια φορά ακόμα εμείς ως χώρα έχουμε μία άποψη, η οποία ενδεχομένω δεν συμβαδίζει με αυτή του Συμβουλίου, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή εκφράζω το Συμβούλιο, γιατί είμαι χώρα τη Μεσογείου. Η Μάλτα, η Ιταλία θα ήθελαν να επενδύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην Βόρεια κυρίως Αφρική και στις όμορες χώρες έτσι ώστε να αποθαρρύνουμε τη μετανάστευση και να τη διαχειριστούμε πριν φτάσει στις ακτές μας. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα ότι οποιαδήποτε επένδυση γίνει εκεί ε, δεν μπορεί να συγκριθεί με την τεράστια απόδοση που θα έχει η επένδυση αυτή για την Ευρώπη από τη μείωση της μετανάστευσης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε το Συμβούλιο και αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, ας το κάνουν οι Εστονοί. Αλλά θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια έτσι ώστε ο φάκελος αυτός να κλείσει και να έχουμε αυτή την εντολή σε επίπεδο ΕΤΕ για εξωτερικό δανεισμό για δανεισμό εκτός ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Εμείς όμως εδώ, επαναλαμβάνω, ε, εκφράζουμε τη θέση του Συμβουλίου. Και για τις χρηματοπιστωτικές οικονομίες και για την αγορά κεφαλαίων πολιτική πολιτική απόφαση για την τιτλοποίηση, το είπε και ο πρόεδρος, όπως επίσης και για τα επενδυτικά κεφάλαια κινδύνου και το Ταμείο για, την κοινωνική, για το κοινωνικό επιχειρήν. Νομίζω ότι ο εισηγητή εδώ για την τυπλοποίηση έκανε καταπληκτική δουλειά. Έδειξε να το έχει το θέμα με τη δική μας βοήθεια και είμαστε πολύ περήφανοι που έκλεισε. Που φαινόταν αδύνατον κάποια στιγμή. Και να σας πω πως προσπαθώντας να ε, επανεκκινήσουμε αυτή την αγορά, να δείτε που θα βρεθούμε και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο το χρειάζονται. Επίσης, τα άλλα δύο ταμεία που είναι του κοινωνικού επιχειρήν και του ε, κεφαλαίου κινδύνου θέλει να δώσει πρόσβαση σε μικρές επιχειρήσεις, σε κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, ανοίγοντά του νέες επενδυτικές δυνατότητες για ταμεία που καλύπτουν μια μεγάλη κλίμακα πιθανών οχημάτων και διαφόρων ειδών διαχείρισης. Οι συνομοθέτης ή συνομοθέτες Επίσης, προχώρησαν πολύ ε, με την οδηγία κατά της, ε, για την νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος και νομίζω ότι αυτά θα, θα μου κάνετε και πολλές σχετικές ερωτήσεις. Να σας πω πως για το τελευταίο θέμα δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα αρκετά που ήταν η καταπολέμηση ε, των ε, παράνομων εσόδων που χρησιμοποιούνται για την τρομοκρατία και για την εγκληματικότητα γενικότερα. Ξέρετε πως ε, εδώ το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ρευστό και το θέμα τελικά είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε σκεφτεί στην αρχή. Παρ' όλα αυτά η Προεδρία της Μάλτας θεωρεί πως ενδεχομένως και το φάκελο αυτό θα τον κλείσουμε και αν έχετε ερωτήσεις με χαρά να απαντήσω. Για να σας πω πως αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο ξανασυζητάμε το θέμα. Στο Συμβούλιο έχουμε ζητήσει να φανούμε πιο ευέλικτοι και να δημοσιοποιούμε ε, τον τελικό ε, ωφελούμενο, να αποκαλύπτεται δηλαδή η ταυτότητά του. Κάναμε επίσης πρόοδο στη συζήτηση Ε, του θέματος της ανάκτησης και της ε, λύσης των ε, Central Parties και να σας πω πως προτείναμε εδώ τη σχετική νομοθεσία που έχει ως σκοπό να κάνει πιο αποδοτικούς και αναλογικούς τους κανόνες που ισχύουν. Και θα προσπαθήσω να κλείσω λέγοντάς σας πως υπάρχει το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης και στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου καταλήξαμε σε μια γενική προσέγγιση για την ιεράρχηση των πιστωτών, όπως επίσης και για τις προτάσεις για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς των υπαριθμών 9. Αυτά. Και αν θέλετε, όταν μου κάνετε ερωτήσεις, μπορώ να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω όμως πως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι η ΟΝΕ έχει ε, ενισχυθεί. Έχουμε κάνει μια εμβάθυση, όπως είπαμε και στη Βαλέτα, τον Απρίλιο. Έχουμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ελπίζουμε ότι και εκεί θα γίνει κάποια πρόοδος όσο περνάει ο χρόνος δεδομένης και της πιο θετικής πολιτικής τάσης που αντιμετωπίζουμε. Τελείωσα λοιπόν και πιστεύω πως γενικά, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε ο τίμιος μεσίτης. Ο τίμιος ενδιάμεσος που άφησε πίσω τα δικά του συμφέροντα και αναφέρθηκε στα θέματα του CMU, την φορολόγηση και στην ε, σχετική νομοθεσία, την οποία πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές πετύχαμε. Ευχαριστώ, Εντουάρ. Πραγματικά ήσασταν ένας έντιμος ε, διαμεσολαβητής, ο κύριος Χέις, πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα και τα συγχαρητήριά μου στην Μαλτέζικη Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε του τελευταίου έξι μήνε. Σε εσά και στην ομάδα σα, και η Μάλτα είναι μικρή χώρα, όπω και η δική μου, οπότε καταλαβαίνω ότι από οργανωτική σκοπιά είναι δύσκολο πράγμα να οργανωθεί μια τέτοια Προεδρία και καλό είναι να το αναγνωρίζουμε. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, μπορείτε να μου πείτε τη δική σας άποψη ως πρόεδρου του ΕΚΟΦΗΝ. Ποια είναι η, γνώμη σας ε, για την πρόταση CCTV. Υπάρχει πλέον μια πρόταση από τον κύριο Μοσκοβισή που προτείνει δύο στάδια. Μια ε, συμφωνία για τη βάση και στη συνέχεια μια φάση για την εξυγίαση. Και όπως γνωρίζετε ε, εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε εξετάσει το θέμα πολύ στενά. Ξέρω ότι τα μεγάλα κράτη-μέλη ε, εκφράζονται πολύ θετικά δημόσια για την πρόταση αυτή, αλλά στους, διαδρά, στους διαδρόμους του ΕΚΟΦΗΜ ε, λένε τα αντίθετα και τηρούν αρνητική στάση. Συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε την ευθύνη για την υποβολή αυτής της πρότασης να συντάξει μια μελέτη επιπτώσεων αναχώρα της πρότασής της καθώς κινούμαστε προς την κατεύθυνση της συμφωνίας και της ε, εξηγήσεις. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο θέμα ως προς τις συζητήσεις που έχετε με τους συναδέλφους σας, τους ομολόγους σας. Και δεύτερον, βάσει του CMU υπήρξε συμφωνία στο θέμα της τιτλοποίησης ε, επί Προεδρίας. Είναι μεγάλο επιτεύγμα αυτό. Όμως, για την τυκλοποίηση τα βύση, όλα αυτά είναι δομικά στοιχεία του CMU. Αλλά ως χώρα που έχετε ιστορικά ε, στενές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η δική μου. Πώς θα λειτουργήσει αυτό ε, στο πλαίσιο του, του Brexit, που έχει την πιο διαφοροποιημένη κεφαλαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς, πώς μπορούμε να λύσουμε αυτόν τον γρίφο σε μια κατάσταση κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκινήσουμε με το δεύτερο ερώτημα και μετά θα, περάσουμε, θα περάσω στο πρώτο. Πολύ σύντομα. Όταν εκλέχθηκα ευρωβουλευτής, είχα έρθει πραγματικά την περίοδο που βρισκόμασταν στο μάτι του κυκλώνα της κρίσης. Ήμασταν οι πιο ε, απασχολημένοι με το μεγαλύτερο, με το πιο επιβαρημένο φορτίο, ε, φόρτο εργασίας επιτροπή λόγω των αρμοδιοτήτων μας. Ήμουν εδώ στην επιτροπή και φυσικά είχαμε, τις, είχαμε εξελίξεις εκείνη την περίοδο. Γεγονός σε κάθε περίπτωση είναι ότι σε τελική ανάλυση βασιζόμαστε υπερβολικά πολύ στις τράπεζες. Και ως ανεπτυγμένες πλέον αγορές χρειαζόμαστε και εναλλακτικέ. Και αυτό είναι θετικό και για τις εταιρείε, οι οποίες έχουν ε, καλύτερους πόρους χρηματοδοτικούς, μακροπρόθεσμους, με καλύτερο επιμερισμό των ε, κινδύνων, παρά του να δανείζονται μόνο από τις τράπεζες. Και είναι ωφέλιμο και για τους ε, καταθέτες, το να έχουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ώστε να επιμερίζονται και οι κίνδυνοι αλλά και τα πλεονεκτήματα, το ωφέλη μια πλήρω λειτουργούσα κεφαλαγορά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Στην Ευρώπη ακόμη δυστυχώ ε, βασιζόμαστε υπερβολικά πολύ στι τράπεζε όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ε, επιχειρήσεων. Χρειάζεται να κινηθούμε σε διάφορες ε, κατευθύνσεις. Τιτλοποίηση, ε, όλες οι άλλες πρωτοβουλίες νομοθετικές. Ε, υπάρχουν τα, τα fintech, τα blockchain, όλα αυτά είναι, είναι, είναι νέοι όροι τους οποίους συζητούμε, αλλά ε, γεγονός είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν και χρειάζεται να αλλάξουμε και νοοτροπία στην Ευρώπη. Να είμαστε πιο θετικοί ε, απέναντι σε άλλες ε, κεφαλαιακές πηγές Φυσικά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι καταθέτες θα έχουν εγγυημένε τι καταθέσει τους. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κινηθούμε στον στο, δρόμο που περιέγραψα. Όσον αφορά το CCCTB και την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Αυτό πρέπει να το εξετάσει κανεί στο ευρύτερο πλαίσιο. Πολλά νομοθετήματα, αναφέρομαι στην ATD1 και ATD2, και λόγω της παγκόσμιας κατάστασης όπου πραγματικά έχουμε μια τεράστια γκάμα ε, κινήσεων από επιχειρήσεις. Ε, πρέπει να τα καλύπτουμε όλα. Το CCCTB είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τι έγινε ε, στο CFC, στο ATADN. Έχουμε δηλαδή θυγατρικές που δεν είχαν αντικείμενο, πλέον θα φορολογούνται. Έχουμε τη διάταξη για το κεφάλαιο εξόδου. Άρα οι εταιρείες πια δεν μπορούν απλά να χρησιμοποιούν ε, τους τόκους για έκπτωση φόρου. Έχουμε τις πατέντες. Όλα αυτά είναι εργαλεία για την Καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η CCTV είναι ένα από αυτά τα εργαλεία. Στις συζητήσεις λοιπόν αυτό που ανέκυψε είναι ότι ε, φάνηκε ότι το εργαλείο αυτό κατα, χαράσει έναν άλλο δρόμο αλλά ε, καταλήγει στον ίδιο στόχο. Υπήρξε λοιπόν το ερώτημα γιατί δεν ακολουθήσαμε τον ίδιο δρόμο. Οι γνώμες διήστανται στο Συμβούλιο. Έχουν υποβληθεί και κάποιες ε, τροποποιήσεις στην πρόταση της Κομισιόν και από την ίδια την Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως Προεδρία εξασφαλίσαμε ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση και θα παραδώσουμε το, το θέμα αυτό στην ε, Εστονική Προεδρία βάσει των όσων ήδη έχουμε επιτύχει εμείς βεβαίως. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, διότι όπως ήταν τα πράγματα κατά την αρχική του φάση τουλάχιστον, προφανώς απέτυχαν, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και εμείς ε, και η Κομισιόν. Κυρία Περές. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι ανήκω σε μια ομάδα που ελπίζει ότι όταν δεν θα πλέον επικεφαλής του ΕΚΟΦΗΝ από την Προεδρία θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε το εγχείρημα αυτό και να μας υποστηρίζετε και εμάς γιατί πρόκειται για ένα εγχείρημα στο οποίο έχει καθυστερήσει περιβολικά η Ευρώπη και στη ζώνη του ευρώ. Βλέπουμε πόσο πολύ χρειάζεται να προχωρήσουμε προς αυτές ε, τις κοινέ ε, διαδικασίες λήψη αποφάσεων, όχι μόνο για να καταπολεμήσουμε το φορολογικό ντάμπινγκ, αλλά και για να προχωρήσουμε προς μια πιο ενιαία βάση φορολογική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα πω, κύριε Υπουργέ, ότι ελπίζουμε να είστε στο πλευρό μας όταν έρθει η ώρα, ακόμα και αν δεν προεδρεύετε του Συμβουλίου. Αναφερθήκατε στο aggregate fiscal stance μεταξύ των καινοτομιών που εισήγαγε η Προεδρία σας. Θέλετε να μου εξηγήσετε λίγο πώς προτείνετε στη συνέχεια να αξιοποιήσουν ε, τη έννοια αυτή οι διαφοροί και σε σχέση με το κοινοβούλιο που χρόνια τώρα το ζητάει. πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη συζήτηση αυτή. Επίσης έχω μια άλλη παρατήρηση για τον φόρο προσθέμενης αξίας, διότι παρατηρώ πως από το τελευταίο κοφήν εκδηλώθηκε μια προσπάθεια εξουδετέρωσης ε, των διεκδικήσεων αφενός της Τσεχίας, αφετέρου της Γαλλίας, σε συνθήκες άθλιες. Και ενώ το Κοινοβούλιο είχε σαφώς ε, υποστηρίξει την ευθυγράμμιση των ε, συντελεστών ΦΠΑ για το βιβλίο, είτε σε ε, έντυπη μορφή, είτε επί χάρτου, δηλαδή είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, εδώ πώς νομίζετε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε αυτή, από αυτήν την κατάσταση. Απάντηση. Κοιτάξτε. Πρόκειται όντως για μια όχι απλώς απογοητευτική, αλλά μια νέα εξέλιξη που δεν είναι καθόλου θετική. Και αν δεν απατώμε, και αρκετά μέλη του Συμβουλίου έκαναν αντίστοιχη παρατήρηση. Εμείς προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τη δυσκολία προτείνοντας τόσες ε, διαβεβαιώσεις σε όρους ε, διασφαλιστικών δικλείδων δηλαδή. Μπορεί να μην ε, παραβλάψουν το σύστημά μας, που είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Αν μια χώρα λοιπόν λέει ότι πιστεύει πως η μεταβολή του συστήματος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης που είναι μεγάλη στη χώρα από ό,τι φαίνεται. Αν και κανείς δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Για χώρα που έχει φορολογικό κενό στα έσοδά τη, δηλαδή είναι μεγάλη η απόκληση μεταξύ αυτών που θα έπρεπε να εισπράττει και αυτών που τελικά εισπράττει. Και είναι μεγάλη και επένδυση, θα πρέπει να δαπανίσουν πολλά χρήματα. Ε, τίθε το ερώτημα πόσο χρόνο τους δίνουμε περιθώριο για να προσαρμοστούν. Πέντε χρόνια, δέκα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν εμείς προτείναμε κάθε χώρα να μπορεί να το εφαρμόζει μέσα στο περιθώριο, μέσα, στο πνεύμα του πρόκειται για γειτονική χώρα. Αλλά δυστυχώς και χωρίς να μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, δεν ήταν η χρονική στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα κατάλληλη για μια τέτοια δοκιμή ή πιλωτικό πρόγραμμα. Όπως είπατε και εσείς ήταν απογοητευτικό αυτό. Και βέβαια κατέστησα φες και τι μας είπαν ότι είχαν κάποια προβλήματα αλλά δεν είναι σχετικά με το e-box. Αυτά τα είχαν δεχτεί. Λοιπόν και έτσι ως ε, Προεδρία αλλά και ω μέλο του Συμβουλίου αναγκαστικά βέβαια και εγώ καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα ότι ήταν απογοητευτικό. Βέβαια για το e-box καταλήγουμε όλοι στο ίδιο, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι κόσμημα, και έχουμε και ένα έγγραφο εργασία για τη διακυβέρνηση αυτή και για το πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Άρα θεωρώ ότι είναι κρεμής η υπόθεση. Από τα σχόλια βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Κάποιοι αποδίδουν ε, ευθύνε στον δικτή 3% για το αν θα πρέπει να υπάρχει ενοποίηση ή αν θα πρέπει να είμαστε πιο θετικοί σχέση με μια σύγκληση άρα με δείκτες που θα δείχνουν ότι υπάρχει σύγκληση χωρών. Ε, όλα αυτά ε, ε, γέρθησαν στο τελευταία συνεδρίες του Συμβουλίου. Και η δική τη δική σας τη δυσφορία τη συμμερίζονται και άλλες χώρες και, άλλα, και μέλη του Συμβουλίου. κύριος Λούκα. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε. Έχετε έναν απολογισμό διατυπώσει για το εξάμεινο της Προεδρίας. Θα ήθελα απλώς ε, να επισημάνω για το εξάμεινο για το οποίο εκφράσετε την ικανοποίηση σας και την κατάσταση του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξή. Γιατί είπατε ότι θεωρείτε πως έχει επιτύχει η Τραπεζική Ένωση. Η Τραπεζική Ένωση και η νομοθεσία που αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα έχει επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και την προστασία του φορολογουμένου σε σχέση με διάσωση τραπεζών. Τώρα όμως βλέπουμε δύο διαδοχικές κρίσεις. Τη Μόντε Ντεϊπάσκι που πάλι χρειάστηκε να διασωθεί με εγγύησεις ε, κρατικές, άρα χρησιμοποιήθηκε χρήμα του Ευρωπαίου φορολογουμένου για τη διάσωση, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε δεν μπορεί να μας ικανοποιεί και την περίπτωση της Μπάνκο Ποπολάρο που δεν διαγνώστηκε ή και αν διαγνώστηκε αντιμετωπίστηκε με τρόπο εσφαλμένο η κρίση. Μια τράπεζα η οποία είχε περάσει επιτυχώς δύο ε, stress test για να καταρρεύσει κάποια στιγμή ξαφνικά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, από όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα, έχει βελτιωθεί κάτι? Έχουμε μπορέσει να καταστήσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα πιο ασφαλή, μπορούν να διαγνωστούν ταχύτερα, πιο έγκαιρα τα προβλήματα. Ή μήπως τελικά και με την εμπειρία που έχουμε αποδεικνύεται ότι ήταν αποτυχημένη αυτή η πολιτική. Απάντηση. Κοιτάξτε, η ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης ε, ε, συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου, της δικής μας Προεδρίας. Μάλιστα ήταν επιδίωξη να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν ταχύτερη, μεγαλύτερη πρόοδο. Για το ίδις τώρα, για την ε, ασφάλιση των καταθέσεων και τα μέτρα περιορισμού του κινδύνου, είχαμε εν γέννη μία συμφωνία για το πρώτο θέμα, ότι θα έπρεπε να εργαστούμε βεβαίως ταχαίως, σε ταχύς ρυθμούς, για την πρόταση. Ταυτόχρονα όμως, δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα στα μέτρα περιορισμού του κινδύνου. Και με ικανοποίηση μπορώ να πω ότι έχει υιοθετήσει δύο γενικές προσεγγίσεις το Συμβούλιο στην προκειμένη υπόθεση με έκθεση προόδου. Και δεν ήταν εύκολο αυτό. Το θέμα, παραδείγμα της χώρας ε, υποδοχής και των λοιπών χωρών ε, ήταν πολύ ευαίσθητο και χρειάστηκε πολύ ενέργεια για να το λύσουμε. Αλλά μπορέσαμε να εξεύρουμε ισορροπία. Οι δε γενικές προσεγγίσεις, η πρόταση σχετική με την ιεραρχία των πιστωτών σε περίπτωση διάσωση μια τράπεζα, που ήταν πολύ σημαντική γιατί όριζε βήμα το βήμα τι πρέπει να γίνει, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και παράγοντα δυσφάλιση των επενδυτών, γιατί θα μπορούσαν έτσι, αν ήταν ομολογιούχοι, να ξέρουν ότι ομόλογα, οι ομολογίες τους θα μετατρέπονταν σε μετοχές και έτσι να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Άρα είχαμε αυτές τι γενικέ προσεγγίσεις, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έχετε με την γνωμοδότηση σα και βέβαια μεταβατικές ρυθμίσεις σε σχέση με το EFRS 9, κεφαλαιοκικές απαιτήσει και συνέπειες και μεγάλη έκθεση. και θα πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει σύντομα. Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει σύντομα τι διαπραγματεύσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Έχουμε, δώσει πολύ, έχουμε κάνει πολλή προσπάθεια όλα τα θεσμικά όργανα ή άλλα όργανα που με κάποιο τρόπο έχουν να αναμειχθούν κάποια στιγμή στην υπόθεση αυτή, έχουν προσκληθεί στη Βαλέτα, χωρίς όμως να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει κάποια εύκολη συνταγή και λύση που θα έλεγε καν αυτό μην κάνεις το άλλο. Και βεβαίως είναι λογικό αυτό, είναι τόσο περίπλοκο το ζήτημα. Τώρα περιμένουμε τις συστάσεις. Έχουν διατυπώσει τις εκθέσεις τους οι εμπειρογνώμονες μας ε, που γραμμίζουν το ζήτημα και προτείνουν λύσεις. και περιμένουμε εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δαλνίων που πιστεύουμε ότι θα πρέπει μέχρι τον Ιούλιο να έχουν υιοθετηθεί. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, αναμονή δηλαδή των εθνικών σχεδίων. Και είχαμε και μια υποομάδα που ξέρετε εργαζόταν εντατικά. Είχαμε την ΕΚΤ με την γνωμοδότησή της. Δηλαδή οι ικανότεροι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και είπαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε έτοιμες συστάσεις για την προσέγγιση του προβλήματος, χωρίς να είναι κάτι το ε, απλό για την... Ε, ναι, αλλά εγώ σας παρακάλεσα να μου σχολιάσετε για την μόντε Monte dei και την ε, Banco Popular. Συμβούλιο δεν έχουμε συγκεκριμένη θέση. Μα τα μέτρα που ίσχυαν δεν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θα έπρεπε κανονικά να έχετε άποψη από, αυτόν τον, από αυτού του θέματος. Όχι. Δεν θα τοποθετηθώ. Πρέπει να δούμε συνολικά τις συστάσεις και δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το Συμβούλιο. φυσικά είναι ε, λογικό ε, το ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου δεν θέλει να ε, τοποθετηθεί για συγκεκριμένες τράπεζες. Προφανώς το θέμα που συζητούμε είναι που υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, και προβλήματα και ο κύριος Λούκ αυτό προφανής να, προφανώς προσπαθεί να τοποθετεί. Αν είχα, λέει ο κύριος Κυκλούνα, άποψη θα σας την έλεγα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άποψη. Ο κύριος Τόιρερ, θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Πρόεδρε, Αναφερθήκατε στις επιτυχίες τη Μαλτέζικη Προεδρία. Θα ήθελα εκ μέρου των φιλελευθέρων και εγώ να δηλώσω ότι είμαστε κι εμεί περιχαρεί που προχώρησε το θέμα της τετλοποίηση έπειτα από έναν επιτυχημένο τριμερή διάλογο όπου αυτό που είχαμε κατά νου ήταν βεβαίως να υποστηριχθεί η πραγματική οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφερθήκατε στην πρόοδο που ε, σημειώθηκε ε, όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, επιθετικής ε, φοροαποφυγής, όσον αφορά την ε, ρύθμιση των υβριδικών δομών ε, ένα, ένα από τα βασικά θέματα ήταν ε, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ανελήφθη σχετική πρωτοβουλία, ωστόσο μας προκαλεί απορία το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατέληξε σε απόφαση προτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ενημερώθηκε αλλά δεν συναποφασίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε την ευκαιρία ούτε καν να ε, γνωμοδοτήσει να καταλήξει στη δική του έκθεση και θα ήθελα να, πω, να εκφράσω την ε, δυσαρέσκειά μας είναι αγενές τουλάχιστον να μην ε, σας ενδιαφέρει η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην την περιλαμβάνετε και να μην την εντάσσετε στη δική σας άποψη. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο το Συμβούλιο δεν περίμενε τουλάχιστον να μάθει την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι η στάση μας ε, θα ήταν, ήταν έτσι κι αλλιώς επικοδομητική. Όσον αφορά την ε, νομοθεσία για την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, περιμένουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, θεωρείτε ότι η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία επαρκεί ώστε να βγαίνουν στη δημοσιότητα εξελίξεις όπως αυτές που είχαμε με τα Panama Papers. Ε, επαρκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να, να αποκλειστούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον ή έχετε σκοπό ε, να αναλάβετε και περισσότερες ε, πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της ε, καταπολέμησης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στο μέλλον. Νομίζω ότι αναφέρεστε στην, στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις διπλής φορολόγησης. Για, για, για τη διπλή φορολόγηση, ναι, το Συμβούλιο έλαβε απόφαση προτού καν προλάβει το Κοινοβούλιο να ε, αποφασίσει, να, να ψηφίσει. Ε, ήταν αγένεια τουλάχιστον αυτό, διότι η στάση μας ήταν πολύ επικοδομητική και νομίζω ότι ο και όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα ήθελε να είχατε λάβει υπόψη σας την δική μας τοποθέτηση. Δεν το γνώριζα αυτό Πάντως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η, έγκριση αυτού θα γίνει μετά την ε, λήψη απόφαση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι πληροφορίε που έχω. Και το δεύτερο ερώτημά μου σχετικά με την νομοθεσία για την καταπολέμηση τη νομοποίηση παράνομων εσόδων Πιστεύετε ότι αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας επαρκούν ή θα προτείνατε η επόμενη Προεδρία να προχωρήσει σε θέσπιση περαιτέρω ε, νομοθετημάτων. Φυσικά περιμένουμε και, άλλ, και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και άλλες νομοθετικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα για τους ενδιάμεσους. Ε, να μην επιτρέπεται δηλαδή ε, σε ιδρύματα χρηματοπιστωτικά να δίνουν συμβουλές που οδηγούν σε επιθετική φοροαποφυγή. Επίσης ε, και όσον αφορά την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα ε, και εκεί αναμένουμε νέα νομοθετικά βήματα. Στη το ίδιο. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα, ε, πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Προς το παρόν έχουμε ολοκληρώσει κάποια βασικά στάδια, αλλά το, η δουλειά αυτή είναι πραγματικά πάρα πολύ ολοκληρωμένη. Χρειάστηκαν χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα και με αυτόν τον τρόπο χαράσει και τον, τον δρόμο που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα. Η νομοθεσία που έχει δημοσιευτεί, που έχει εγκριθεί ε, μέχρι στιγμής, δεν έχει τεθεί ακόμη πλήρως σε εφαρμογή. Μόνο τότε, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείε επενδύουν, μετακινούν, μεταφέρουν κεφάλαια κτλ. Πέραν αυτών, βάσει, ε, ε, αυτές είναι υποχρεώσεις που απορρέουν και από τον ε, ΟΣΑ. Είμαστε και στο παγκόσμιο επίπεδο ε, υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε ηγετική θέση μάλιστα, ώστε όχι μόνο εμείς αλλά και οι τρίτες χώρες να προχωρήσουν σε αλλαγές. Θυμάστε και τον κώδικα διοντολογίας ε, όσον αφορά την, ε, την κατονομασία και την, των, των, των χωρών που δεν θα υιοθετήσουν τις ελάχιστες απαιτήσει που έχουμε εμείς στην Ευρώπη για τις φορολογικές αρχές και την υποβολή εκθέσεων αναχώρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η δημοσίευση αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι αρχές των χωρών έχουν πλέον πολλές πληροφορίες και αρμοδιότητες πρώτον για να ανταλλάσσουν πληροφορίες για παράδειγμα για τις αποφάσεις tax rulings υπάρχει πλέον από, ε, απόφαση, υποχρέωση κάθε φορολογική αρχή να ε, κοινοποιεί ε, με, στις άλλες 27 φορολογικές αρχές τυχόν τέτοιες αποφάσεις που λαμβάνει. Αυτά είναι μέτρα που νομίζω ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σημαντικά στον τομέα αυτό. Το πρόβλημα δεν αφορά τη δική σας Προεδρία. Αφορά γενικά το Συμβούλιο. Πολύ, το Συμβούλιο πολύ συχνά υιοθετείται ε, γενική προσέγγιση προτού ε, καταφέρουμε εμείς να τοποθετηθούμε. Δεν, δεν μας ακούτε και νομίζω ότι αυτό μπορεί να ακολουθεί το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα των ε, συνθήκων. Κυρία Κάπελ, ευχαριστώ πολύ. Τρία θέματα θέλω να θέσω. Πρώτον, καταπολέμηση φοροαποφυγής. Ένα θέμα με το οποίο ασχολείται η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το τελευταίο εξάμεινο. Ε, συζητήθηκαν και διάφορα θέματα. Είπατε ότι επιτύχατε σε δύο τρόπους. Ε, πρώτον στην επίλυση διαφορών στην διπλή και ε, στις, στα, στις χώρες που δεν συνεργάζονται. Ε, τώρα θα ήθελα να θέσω εγώ ένα θέμα στην, ε, στην ε, απάτη ΦΠΑ, για παράδειγμα. Ε, ποιες θεωρείτε, ποιοι, ποιες θεωρείτε ότι, ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι τομεί στην επόμενη πρόεδρε μπορούμε να καταλήξουμε σε, σε, τα αποτελέσματα. Δεύτερο, Ελλάδα. Υπήρξε μια συμφωνία για την εκταμίευση, αλλά όχι για το χρέος και την συμμετοχή του Δουνουτού. Ε, γιατί δεν υπήρξε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί η οποία δεν αναλαμβάνει την αγορά ελληνικών ομολόγων. Ε, επίσης, ε, Σημαντικοί οικονομολόγοι αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα εξακολουθεί να παρακολουθεί τις διαδικασίες, να μην κάνει ό,τι χρειάζεται για την ανάκαμψη της οικονομίας, ότι υπόσχεται πολλά αλλά δεν υλοποιεί πολλά. Μεσοπρόθεσμα το Συμβούλιο όσον αφορά την βιωσιμότητα του χρέους της, της Ελλάδας θα ε, καταλήξει τελικά η διαδικασία αυτή σε κούρεμα ή το Συμβούλιο έχει μια άλλη στρατηγική. Όσον αφορά το έγγραφο προβληματισμού για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της ΟΝΕ, το ΕΚΟΦΗΝ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την παροχή ε, κινήτρων για την υλοποίηση των ε, συστάσεων αναχώρα. Το Συμβούλιο έχει κάποια ιδέα, κάποιο, κάποιο σχέδιο για το πώς μπορούν ε, οι χώρες να οδηγήσουν σε μια ε, πιο εναρμονισμένη φορολογική πολιτική στην Ευρωζώνη. Πολλά... Πολλές ερωτήσεις τυπώθηκαν. Για να δούμε τη σειρά. το ίδιο στα Eurobond, όπως θέλετε πείτε το, το pooling, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά προσκρούν στο ζήτημα του μικρότερου κινδύνου. Άρα, η αδίποτε επιλογή, επιλογή θα βρεθεί ενώπιον αυτού του ζητήματος. Δεν λέω ότι είναι τείχος, αλλά πάντως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Οι χώρες πιστωτές. Γερμανία είναι αυτή, Μάλτα είναι αυτή, όποια χώρα είναι πιστωτής, ή εν περιπτώσει μια χώρα που δεν έχει προβλήματα, θέλει όταν ε, προβαίνει σε εκδήλωση αλληλεγγύης να δει από την άλλη χώρα ότι και η ίδια κινεί τη χείρα της. Με την Ελλάδα, παραδείγματι, που λέτε ότι κάποιοι λένε πως δεν ε, πράττει τα απαραίτητα, βάση περιπτώσει δεν το κρίνω αυτό. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία. Θα σε βοηθήσουμε αλλά και εσύ να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Συνεργασία λοιπόν από χώρε πιστωτέ σε αμοιβαιοποίηση ή κάποιο τύπου εναρμόνιση δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτή την περίπτωση. Για την Ελλάδα η κατάσταση έχει όπως έχει επειδή δεν εκταμιεύονται δόσεις, όπως είπατε, αν δεν αποδειχθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι. Οι όροι ορίζονται για να βοηθηθεί μια χώρα να βοηθήσει τον εαυτό της, να μην χαθούν τα χρήματα, αλλά να αξιοποιηθούν ώστε να στηριχθεί η χώρα, να σταθεί στα πόδια της, να γίνει πιο εύρωστη οικονομικά, να βγει στις αγορές. Αυτή είναι η ελπίδα. Τώρα βέβαια επικρέμαται το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους. Οι δε θέσεις του Δουνουτού διαφέρουν από αυτές των Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το σημαντικό λόγο. Και γι' αυτό και επειδή η Ελλάδα είναι μέλο τη οικογένειά μα μακροπρόθεσμα, έχουμε διαφορετικού κανόνε. Βέβαια, το Δουνουτού έχει διαφορετικού κανόνε ε, που είναι υποχρεωμένο και να τηρεί, διαφορετικού από του δικού μα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δράσουμε από την απαραίτητο, από την αιτιολογημένο, με μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, όχι απαραίτητο όμως με κούρεμα. Μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι, γιατί Μάλτα θα δώσω ένα παράδειγμα, που ε, δανείζεται χρήματα σε, ποσοστό υψηλό, σε επιτόκιο υψηλότερο από αυτό που δίνει στην Ελλάδα ή παίρνει από την Ελλάδα όταν τις δανείζει. Αλλά αυτό είναι η ελληνική. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε το χρέος να μην είναι βάρος για τη χώρα. Αλλά όχι βέβαια κούρεμα. Πάντως, στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Διεθνές Σωματικό Ταμείο καταρχήν, καταρχήν συμφώνησαν και βέβαια τώρα πια επιστρέφει η πρόεδρος του Διεθνού Σωματικού Ταμείου στο Συμβούλιο, το διοικητικό, αλλά από την άλλη και εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά και τις δικές μας εκτιμήσεις και φαίνεται ότι έχουμε καταρχήν τουλάχιστον βρει ε, έναν τρόπο συμβίωσης με τους, μέσα στους όρους που έχουμε ορίσει. Ευχαριστώ πολύ και τώρα πρέπει να ομοδοποιηθούν οι ερωτήσεις γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη θέση μας με τη διερμηνία. Παρακαλώ λοιπόν να ακούσουμε με τη σειρά ο κύριος Λάγκεν. Ναι, πάντως εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είπατε και το σημείωσα ότι η καταπολέμηση της νομοποίησης παρανόμων εσόδων είναι δύσκολο ζήτημα. Έχει ε, ε, περιπλακεί ακόμη περισσότερο λόγο της υπόθεσης των εγγράφων του Παναμά. Το συζήτησαμε και έχετε δίκιο σε αυτό το σύστημα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Μας είπε ο Υπουργός ότι, ο Πρωθυπουργός ότι έχετε τέσσερις εκκρεμείς ε, έρευνες, εκτός, ε, μεταξύ των οποίων υπάρχει και μια που αφορά την ίδια τη γυναίκα σας. Αλλά μόνο αυτή έχει σχέση με τα έγγραφα του Παναμά. Άλλε τρει που δεν έχουν σχέση με το Παναμά επίση είναι εξέλιξη. Και θα θυμάστε κι εσεί προσωπικώ από το Fact Finding Mission που είχαμε στην ε, Μάλτα, την αποστολή την ε, διαρευνητική και μιλήσαμε με τι αρχές αλλά και με εσά τον ίδιο γιατί ήταν σε ένα μέρο τη αποστολή μα παρόν ε, όπου υπόθηκε ότι οι έρευνες κατά μέλλον της κυβέρνησης και ο κύριος Μίτση ε, ανέλαβε ακόμη πιο σημαντικά τώρα καθήκοντα για την κυβέρνηση της, Μάλκα, της Μάλτας. Ε, εν πάση περιπτώσει, οι αρχές ε, οικονομικές ε, δίωξης οικονομικών εγκλημάτων υποβάλλουν στον πρόεδρο ή στον διοικητή της αστυνομίας σχετικά αιτήματα, ο οποίος βλέπουμε εντωμεταξύ να έχει παραιτηθεί, και ο διαδοχός του λέει «Α, δεν κάνω τίποτα με αυτές τις καταγγελίες αν δεν αναλάβει δράση δικαστή. Γιατί τα λέω αυτά. Γιατί παρακολουθώ και από το Facebook και από τα μέσα μαζική ενημέρωση, τον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοί του ΕΛΚ, οι κύριοι Κάζα και Μετσόλα, αντιδρούν στην υπόθεση των εγγράφων του Παναμά και καταγγέλουν τους εχθρούς της Μάλτας. Είναι δυνατόν. Εν πάση υπάρχουν και κάποιοι φίλοι της Μάλτας και στη Μάλτα και ο Αρχιεπίσκοπος που είναι ε, καθολικός ιερέας ε, αυστηρών αρχών και με αυτό θέλει να τηρήσει τους όρους. Μα, όχι θα με ακούσετε γιατί δύο φορές έχω γραφεί τους ε, δημοκρατικούς κανόνες. Λοιπόν, έχω τα εξή να ρωτήσω. Πρώτον, ε, ξεκινούν τέτοιε έρευνες και ανακρίσεις ή έχουμε μείνει στην κατάσταση του τέλους Φεβρουαρίου ότι δηλαδή το σπρώχνουμε όλο κάτω από το χαλί. Και για σας ναι, θα πω ότι έχετε κάνει καλή δουλειά, καμία αμφιβολία, σας ε, πάντα γι' αυτό. Αλλά, αλλά η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης ή ενός μέλους της ε, πάβει εκεί που δεν είναι ειλικρινής και έντιμος ή έντιμη. Για τον κώδικα συμπεριφοράς. Έχουν απαντήσει τα 20 κράτη-μέλη, εσείς όχι. Πρόκειται για ένα διακυβερνητικό εργαλείο, όπου λογοκρίνονται και τα έγγραφα. Επομένως, γιατί δεν απαντάτε. Και μπαίνει μέσα σε μια μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων η Μάλτα, που από ό,τι φαίνεται και από πληροφορίες που έχουμε, αν κανείς πληρώσει 35% φόρο επί των ε, εισοδημάτων κάποιους του κάνουν επιστροφή φόρου 30%. Μα όχι, ε, το ξέρω πρόεδρε, το ίδιο βλέπουμε κάθε φορά. Όσοι καταρχάς φρόντισα να καθυστερήσει η εκκίνηση της συνεδρίας κατά μισή ώρα και επίσης όταν έχουμε υπουργό Σαλδημοκράτη και τον ε, ενοχλούν οι ερωτήσεις, τον διακόπτεται τον ερωτώντα. Είχατε δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρος, ξανά, ο κύριος Μοργάνου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις σύντομα. Πρώτον, τέλη Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το έγγραφο αναλογισμού για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση όπου πέραν ε, του πώς έγινε δεκτό, ποια ήταν η ανταπόκριση στο έγγραφο αυτό, στο οποίο απαντήσατε ήδη με προηγούμενη ερώτηση, δεν θέλω να ρωτήσω αν ε, διαπιστώνεται πολιτική βούληση από πλευρά των κρατών μελών για ανάληψη μιας πιο αποφασιστικής πορείας προς την ολοκλήρωση της, της Οικονομικής Ένωσης. Και θέλω ε, να σημειώσω κλείνοντας αυτό το κομμάτι ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας είπε τον Ιανουάριο του 2017 ότι αισθάνεται αμηχανία σε σχέση με την επιλογή ασφαλών ε, ή διασφαλισμένου ενεργητικού. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως εναλλακτική στο ευρωομόλογο. Λοιπόν, δεν θέλω να το σχολιάσω εδώ. Δεύτερη ερώτηση για τις δύο οδηγίες. CCTB και CCCTB. Ήδη δώσατε κάποια απάντηση ενδεικτική προς την κυρία Μπέρες. Θέλω όμως να αντιληφθώ εάν θεωρείται πιθανόν ή αν πιθανολογείται δεδομένων και των εξελίξεων ότι μεταξύ τα κρατών μελών μπορεί να προκύψει δυνατότητα ε, να σχεδιαστεί η απόδοση αυτού του συστήματος ως ε, μερική έστω χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τη μορφή των ιδιών πόρων. Και τρίτον, για τα ηλεκτρονικά βιβλία, δώσατε κάποια ανεκτική απάντηση πάλι, αλλά δεν θεωρείτε ότι μπορεί να αποκόπει το ζήτημα του ΦΠΑ στα βιβλία επί χάρτου και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αφού ε, ούτως ή άλλως πιέζει ο χρόνος, ευχαριστώ Μαρτουσέλο. Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Δύο ερωτήσει. Η Μάλτα ξέρουμε ότι έχει μετατραπεί σε αγαπημένο προορισμό των Ιταλών που μετατοπίζουν τις επαγγελματικές τους, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ε, και το θαύμα αυτό έχει μόνο, μία, μόνο ένα όνομα, ε, απόκρυψη από τα τέσσερα δις εισοδήματος, κάθε τέσσερα δις εισοδήματος αποκρύπτονται σε σχέση με τα άλλα κράτη ε, σημαντικά ποσοστά ποσών που περνούν μέσα από δραστηριότητες, θα έλεγα όχι απολύτως νομότυπες. Ερωτώ λοιπόν, τι, είδους, ε, τι, τι ποσά είναι αυτά καταρχάς, τι ποσοστά είναι αυτά πρώτον και δεύτερον τι μηχανισμοί αναπτύσσονται από τη Μάλτα για την επιβεβαίωση, την ε, ε, επιβεβαίωση της ταυτότητας των ε, επενδυτών και οικονομικών παραγόντων που αναπτύσσουν τις δραστηριότητε τους στην Μάλτα. Επίσης λέγεται ότι θα πρέπει να προσληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι λογιστές πρέπει να έρθουν λέει, να δουλέψουν στη Μάλτα και αν αυτοί δραστηριοποιούνται στη Μάλτα, Ιταλοί, λογιστές και φοροτεχνικοί, ε, λέγεται ότι θα πρέπει να τους καλέσουν και τα επιμελητήριά τους ε, να λογοδοτήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα, με τη συζήτηση που έγινε στο ΕΚΟΦΗΝ, στην ομάδα ενισχυμένες ε, συνεργασίας, το FTT, που δεν ήταν προτεραιότητα δική σας, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω πώς τρέχουν εκεί οι διαπραγματεύσεις. Και δεύτερον, Κάτι που είπα προηγουμένως και θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Στην εγγύηση καταθέσεων ξέρουμε πως το Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο και ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα γίνει και η πολιτική συζήτηση. Οπότε πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, πώς πάει η συζήτηση αυτές τις εβδομάδες. Είμαστε αισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε εξηγήσω πως εδώ έχω έρθει ως πρόεδρος του Συμβουλίου. Δεν είναι προσωπική άποψη. Αυτή η οποία εκφράζω εδώ είναι η άποψη του Συμβουλίου. Γίνεται δουλειά, έχουμε αποτελέσματα, έχουμε προτάσεις, οπότε το μόνο που μπορώ να απαντήσω είναι οι σχετικές ερωτήσεις για τα υπόλοιπα. Βέρνερ, μα εσύ ρώτησες τόσα πολλά. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Όπως έκανα και, στον, ε, και στη Μάλτα και για τα Panama Papers και για όλα και για όλες τις που έκανες. Όμως, τώρα για το νομικό πρόβλημα μεταξύ Συμβουλίου και Παναμά, τα θέματα αυτά είναι υπερβολικά περίπλοκα για μένα. Πάντως, Είμαι υπουργό Οικονομικών τη Μάλτα και γι' αυτό όποτε με καλέσεις μπορώ να έρθω όσε φορές θέλεις και να σου απαντήσω όλες τι ερωτήσεις αυτές. Για το κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση για εμβάθυνση της ΟΝΕ, πιστεύω πως ναι γιατί το πολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή μεταλλάσσεται, όλοι το βλέπουν. Είναι η Γαλλία, είναι άλλα θέματα. Είμαστε στην, μετά τον Brexit ή μετά τον Τραμπ εποχή. Τι να σας πω, πάντως αλλάζει. Και οι πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία αλλάζουν ακόμα περισσότερο το είδο της συζήτηση που κάνουμε στο Συμβούλιο. Δηλαδή είναι πολύ πιο θετικές. Με την έννοια του οράματος, της βούλησης να δράσουμε και αυτή είναι η εντύπωση που μας δημιουργείται. Και ενδεχομένως αυτά θα ενισχυθούν και μετά τις εκλογές. Το κενό και οι αργοί ρυθμοί των εξελίξεων στην ενιαία αγορά αυτή τη στιγμή μοιάζουν, όπως το βλέπω εγώ, και από ό,τι ακούμε στο Συμβούλιο να έχουν ξεπεραστεί και να έχουμε μια αλλαγή προς το καλύτερο, με περισσότερη θέληση για να κάνουμε πιο πολλά. Τώρα, για τα φορολογικά θέματα με την Ιταλία. Εμείς είμαστε σε επαφή με τους Ιταλούς ομολόγους μας, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, σημειώσεις. Για όλα. Τώρα, για λιμένα καταφυγής και για φορολογικό παράδεισο, εγώ μπορώ να φτιάξω ό,τι η ιστορία θέλετε στο μυαλό μου. Δεν είναι ο τρόπος αυτός για να προχωρήσουμε. Υπάρχουν θεσμοί που πρέπει να ενισχυθούν. Και χρειαζόμαστε την ομοθεσία που υπάρχει με την αυτόματη, αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών. Και από εδώ και πέρα θα ισχύσει αυτό κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν και αυτό είναι καθησυχαστικό. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κατηγορεί κανείς ένα μη κλασικό φορολογικό σύστημα γιατί το ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η DG Competition. Και όσα. Εντάξει, σας μπορεί να μην σας αρέσει. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να φτιάχνει κανείς τέτοιου είδους ιστορίες. Τουλάχιστον οι υπερογνώμονες θα έπρεπε από όπου και να προέρχονται τι ακριβώ συμβαίνει και δεν υπάρχει καμία τεκμερίωση στου οποίου να βασίζονται οι παρουσιάσει για το είδε. Μας είπα να συνεχίσουμε τη δουλειά μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, συστατικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης και θα αντιμετωπίσουμε πολλές πιέσεις από παντού. Για να το πετύχουμε. Και το τριπλό CTB με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε τη μετατόπιση κερδών μέσω της μεταφοράς ε, ε, μηχανισμού πληρωμής. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε ακολουθήσει μία τριπλή προσέγγιση. Και πιστεύω πως για το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε συναντήθηκα μόνο μία φορά υπό τη δική μας προεδρία και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Πρέπει να κλείσουμε. Άρα λοιπόν συμπερασματικά θα σας πω πώς οι προσδοκίες δεν ήταν ψηλέ, μικρή χώρα και τα διάφορα, αλλά νομίζω πως αν εξετάσει κανείς τα αποτελέσματά μας, και ελπίζω και μέχρι τα τέλη του μήνα, θα καταφέρουμε να κλείσουμε και μερικά ακόμα, οπότε νομίζω πως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όσα πετύχαμε ως Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πολύ πετυχημένη συνεργασία, για τα εξαιρετικά αποτελέσματα του εξαμήνου που ακόμα δεν έχει λήξει, οπότε κάτι ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε τις επόμενες ημέρες και μετά θα συνεχίσουμε να σας έχουμε εδώ μια και θα είστε ένα τακτικό μέλος του ΕΚΟΦΗΝ και σίγουρα θα συνεργαστούμε θαυμάσια και στο μέλλον. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά που ήρθατε γιατί ήσασταν και αξιότιμο μέλος αυτής της Επιτροπής στο παρελθόν. Γεια σας.